Dear colleagues, can I ask you to take your seats? We will... παρακαλώ, καθίστε. Θα ξεκινήσουμε την ακρόασή μας. Είναι χαρά μου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, να υποδεχτώ την υποψήφια Επίτροπο, την κυρία Σιλβί Γκουλάρ, και δίπλα μου η Συμπρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, της ΙΤΡΕ, θα συμπροεδρεύσει μαζί μου σε αυτή την ακρόαση. Είναι κοινή η ακρόασή μας, όπως τα γνωρίζετε, και επίσης θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Γιούρι και Καλτ, των ε, συνεργαζομένων επιτροπών, καθώς και των Τραν και της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ, που είναι προσκεκλημένες σε αυτή την ακρόαση επιτροπές. Είναι εν είδη εισαγωγής, σαφές από την πλευρά της ΣΥΜΚΟ, ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας είμαστε υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και των μέτρων για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ενδεχόμενων φραγμών για την ε, καλή λειτουργία της ε, εσωτερικής αγοράς επιγραμμικά και όχι και για την προστασία των καταναλωτών από την άποψη της πολιτικής και της νομοθεσίας για την υλοποίηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των καταναλωτών. Γι' αυτό αδειμονούμε για την ακρόαση αυτή για να κατανοήσουμε καλύτερα την προσέγγιση που θέλει να ακολουθήσει η κυρία Γκουλάρ σε σχέση με τα θέματα αυτά, καθώς και για να μάθουμε καλύτερα πώς η υποψήφια επιτροπός σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα ανακύψουν σε αυτό το χώρο. Να θυμίσω ότι η εσωτερική αγορά για τα αγαθά και τι ωφελεί Ιδιαίτερο στους καταναλωτές και τις εταιρείες αρκεί οι κανόνες να εφαρμόζονται κατά τρόπο ισοδύναμο και ισότιμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την εσωτερική αγορά, αποφεύγοντας τον κατακαιρματισμό και τις τεχνητές, τους τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ των νέων ψηφιακών αγορών και των παραδοσιακότερων, για να διασφαλίσουμε ότι οι υπάρχοντες κανόνες είναι εγκαίρος σε θέση να εφαρμοστούν και να γίνουν σεβαστοί. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι σε αυτό το πλαίσιο η, ο τομέας των υπηρεσιών, των υπηρεσιών σε όλες τις ε, διαστάσεις είναι θεμελιώδους σημασία για την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ε, ε, ανάπτυξη, καθώς και την καλή διαβίωση των καταναλωτών στι σημερινέ παγκοσμιωμένε αγορέ. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η νομοθεσία μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, σε κατάσταση επικαιροποιημένη για να αντιμετωπίσει τι προκλήσει του μέλλοντο και να μπορέσουμε και να ε, αντλήσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα καθώ και την ε, μέγιστη δυνατή τεχνολογική πρόοδο. Προστατεύοντα του καταναλωτέ και δημιουργώντα ένα ισότιμο πεδίο για ανταγωνισμό για τις εταιρείε. Ελπίζω ότι θα καταλαβαίνει η υποψήφια Επίτροπο τι μέρημνέ μα για τι μελλοντικέ εξελίξει στην εσωτερική αγορά και την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην εύρωστη, εύρυθμη μέλλον λειτουργία τη και να αντλήσουν τα μέγιστα δυνατά ωφέλη επιχειρήσει, καταναλωτέ και εργαζόμενοι. Κατόπιν αυτών, να δώσω ευχαρίστω το λόγο στην κυρία Βαλέαν τη Επιτροπή Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντεσούτερ. Καλώ ήρθατε όλοι Επιτροπές Ήτρε και ΕΜΚΟ. Θερμό όρισμα και στην κυρία Γκουλάρ που ήρθε ε, για να απευθυνθεί στις δύο επιτροπές μας και για όλους που μας ακούνε και σε αυτή την αίθουσα και από το διαδίκτυο, διότι μεταδίδεται και στο διαδίκτυο αυτή η συνεδρίαση. Να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή Ήτρα είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για ένα τεράστιο τμήμα του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων της κυρίας Γκουλάρ. Βιομηχανική, πολιτική, νέες τεχνολογίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διάστημα, ε, κοινωνία της πληροφορικής, των πληροφοριών, της τεχνολογίας, των δικτύων και των υπηρεσιών. Η ακρόαση αυτή είναι άκρο σημαντική για τα μέλη της επιτροπή μα, διότι το χαρτοφυλάκιο αυτό για μα αποτελεί το πραγματικό μέλλον τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Η ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη, οι μελλοντικέ εξελίξει και οι νέε τεχνολογίε είναι καθοριστικέ. Γι' αυτό, κυρία Γκουλάρ, ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσά τι απόψει σα για το θέμα αυτό. Και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω πώς θα διεξαχθεί αυτή η ακρόαση. Θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγική ομιλία 15 λεπτών από την κυρία Γκουλάρ. Μετά θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από τις εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και κατόπιν «18 ερωτήσεις» οι οποίες έχουν ε, διαιρεθεί μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων ως προς το χρόνο βάσει του συστήματος ΔΕΟΝΤ. Η κυρία Γκουλάρ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να κάνει μια καταληκτική παρέμβαση 5 λεπτών. Τώρα, η διάρθρωση μια ερώτηση ε, και τη απάντησή τη έχει ω εξή. Ένα λεπτό για να θέσει κανεί την ερώτηση και δύο λεπτά για την κυρία Γκουλάρ για να απαντήσει. Και έπειτα, δυνατότητα επερώτηση ενό λεπτού και απάντηση ε, δεύτερη απάντηση ενό λεπτού. Δηλαδή, όριο συνολικό πέντε λεπτά. Ένα ε, για την πρώτη ερώτηση, δύο για την πρώτη απάντηση, ένα και ένα για τις δεύτερες ερωτήσεις και απαντήσεις η επερώτηση καλό θα να αφορά το ίδιο θέμα με την αρχική. Οπότε παρακαλώ μην αποκλίνετε πάρα πολύ, μην κάνετε μεγάλες παρεκβάσεις. Και δουλειά μας εδώ, δική μου και της κυρίας Δεσούτερ, είναι να τηρήσουμε και την ε, ώρα, τα χρονικά όρια. Παρακαλώ λοιπόν να είστε συνοπτικοί όταν θέτετε ερωτήσεις διότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπως το σφυρί ή το να κόβουμε με τα κουμπιά τα μικρόφωνα. Κατόπιν τούτον, να ξεκινήσουμε την ακρόασή μας με, τα 15 λεπτά εισαγωγής από την κυρία Γκουλάρ. Έχετε το λόγο. Κυρίες Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, για όσους μας ακούν από μακριά χάρη στι νέε τεχνολογίες. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση και χαρά που βρίσκομαι εδώ, γιατί έχω πολλές αναμνήσεις από την αίθουσα αυτή και πολλά οικία πρόσωπα που εκτιμώ ιδιαίτερως. Για την επόμενη πενταετία θα ήθελα να δώσω στις ε, επερχόμενες γενιές τα μέσα για να ζουν με βάση τις επιλογές τους, να κρατήσουν, να διαφυλάξουν την κυριαρχία τους. Έναν αβέβαιο κόσμο, η διαφύλαξη των ελευθεριών μας, τη ευημερία μας, του κοινωνικού μας μοντέλου, εξαρτώνται από την ικανότητά μας να φέρουμε σε αίσιο πέρα στην οικολογική μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτές είναι οι δύο κορυφαίε προτεραιότητε και της ε, εκλεγή σα Προέδρου Φοντερ Λάινερ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο χάρτη πορείας και έρχομαι με μεγάλη ταπεινοφροσύνη εδώ για να σας παρουσιάσω κάποια περίπλοκα θέματα για τα οποία είστε περισσότερο ειδήμονες από μένα. Έχω όμω ε, ένα ολόκληρο επιτελείο και ευχαριστώ και το διοικητικό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώ για τη βοήθειά τους και θα βάλω τα δυνατά μου. Καταρχήν, για το δικό μου τομέα, έχουμε πέντε απαιτήσει. Η πρώτη την υπεθύμησε πριν από λίγο ή πρόεδρο ή ή Συμπρόεδρη, Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το δυναμικό τη ενιαία αγορά. Βέβαια θα μου πείτε, α ναι, αυτά το έχουμε ακούσει, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά. Αλλά είναι το απαραίτητο προαπαιτούμενο για την ανταγωνιστικότητα και τις θέσει απασχόληση. Και ενθαρρύνομαι από το γεγονό ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των Brexit κρατήσαμε την ενότητά μα, διαφυλάξαμε το ενιαίο μα μέτωπο υπέρ τη ενιαία αγορά που φτιάξαμε από κοινού. Και μάλιστα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το, και το Κοινοβούλιο να ακολουθήσουν αυτή την πορεία. Οπότε θα ακολουθήσω αυτή την έκκληση. Θα πρέπει επίση να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό των οικονομιών μα. Γιατί μόνο αν έχουμε νέα οικονομική ε, η πυρωτική πολιτική θα βρεθούμε στο απειρόβλητο των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Βέβαια, το να πετύχουμε συνένεση δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί υπάρχουν κάποιε εύλογε προσδοκίε και εκείνων που θα ήθελαν περισσότερου ε, κανόνε και άλλου που θεωρούν ότι είναι υπερβολικοί. Θέλουμε επιστηστική ασφάλεια, κυβερνοασφάλεια, οικολογική ασφάλεια, αλλά και λιγότερε διατάξει για να μπορούν εύρυθμα να λειτουργούν οι επιχειρήσει. Και θα πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε το θέμα των υπηρεσιών ε, βλέπουμε και στη βιομηχανία και στη γεωργία ότι τα όρια μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών είναι πιο ρευστά. Και για να απαντήσω στους επικριτές, πιστεύω ότι για να προσπίσουμε την αγορά μας θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στους επικριτές για την έλλειψη κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης. Η σε Επίτροπος θέλει να συμφιλιώσει την αγορά με το κοινωνικό τομέα. Και γι' αυτό θα ασχοληθούμε με σημαντικά θέματα. Τη θέσπιση ενός ε, δίκαιου κατώτατου μισθού, ε, κοινή ενοποιημένη βάση για τη φορολογία επιχειρήσεων. Μάλιστα ήμουν και συγγήτρια για το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Ε, επίσης, ε, φορολογία των ε, τεχνολογικών γιγάντων, των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Και θα πρέπει να δούμε και τα θέματα των πλατφορμών στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, θα προσπαθήσω αμερόληπτα να φροντίσω για την εφαρμογή των υπαρχών των κανόνων, χάρη σε ε, αυστηρή παρακολούθηση των παραβιάσεων υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα επιβραδύνω λίγο γιατί φοβάμαι πω δεν με παρακολουθούν οι διερμήνε, του οποίου εμπαρόδο ευχαριστώ για το έργο του. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όσοι με θυμούνται από την Επιτροπή ΕΚΟΝ για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη μπορούν να είναι ήσυχοι. Θα φροντίσω ώστε με τα μέσα που έχουμε να εφαρμοστούν οι κανόνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεύτερη απέτηση. Μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα ήθελα μαζί του, αν μου δώσετε την εμπιστοσύνη σα, να είμαι απέναντι στι μικρομεσαίε επιχειρήσει ε, ρεαλιστική. Και όταν ρωτάω τη γνώμη του, μα λένε θέλουμε κατάλληλη στρατηγική, προς, προσβάσιμη χρηματοδότηση, ειδικευμένο προσωπικό, λιγότερη γραφειοκρατία και δυνατότητα να πληρώσουν όταν έχουν ε, ε, χρέη. Επίσης, ε, Έχουμε και το πρόγραμμα InvestEU, αλλά και υπηρεσίε όπω το Solvit για την επίλυση των διαφορών στην ενιαία αγορά, που διευκολύνουν το την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ταμείο Άμυνα. Αυτό είναι μία από τι αποστολέ που μου ανέθεσε η εκλεγήσα πρόεδρο. Θέλουμε επίση να διευκολύνουμε τη συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με του μεγάλου ομίλου και να τους δώσουμε πρόσβαση στη διασυνοριακή συνεργασία για να ανακτήσουν ένα τμήμα τα 10 δισεκατομμύρια ετήσεων επενδύσεων στον τομέα αυτό. Με σεβασμό φυσικά της ε, αρμοδιότητας των κρατών μελών, αλλά και με καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων που έχουν για την ασφάλεια. Και επίσης να πιάνουν τα χρήματα των φορολογουμένων, να έχουμε λιγότερε δαπάνε, αλλά και να έχουμε κατάλληλε στρατιωτικέ δαπάνε όλες οι συνέργειες θα αξιοποιηθούν και για τις τεχνολογίες άμυνας και του μη στρατιωτικού τομέα, κάποια υλικά που θα χρειαστούν για τις μεταφορές, μεταξύ του διαστήματος και της άμυνας, γιατί είπατε ότι η διαστημική πολιτική που ενδιαφέρει την Ήτρε είναι επίση πολύ σημαντική και επίσης διευκόλυνση της κινητικότητας και της στρατιωτικής κινητικότητας. Θέλουμε μια κοινή στρατηγική για την βιομηχανία. Δεν πρέπει να ερθριάζουμε για την οικονομία μα, τι επιδόσει τη, την ευρηματικότητά τη. Άλλωστε, παρέχει το 1 τέταρτο των θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Βέβαια, θα πρέπει η βιομηχανία μα να μεταμορφωθεί άρδιν. Επίση, η κυκλική οικονομία ακούγεται αφηρημένη έννοια. Φαντάζομαι και εσείς θα σοκάρεστε όταν βλέπετε πόσες συσκευασίες έχουμε, πόσα πλαστικά, δεν έχουμε καλή διαχείριση των αποβλήτων, υπάρχει κατασπατάληση τροφίμων. Επίσης, ε, θα πρέπει να βελτιώσουμε τους τρόπους παραγωγής μας, να γίνουν πιο φιλοπεριβαλλοντικοί και να εξοικονομήσουμε πόρους σπάνιων γεών, κάποιων ε, πρώτων υλών που εισάγουμε και να διασφαλίσουμε και την βιοπικιλότητα έχω συνέστηση και το λέω με κάθε ταπεινοφροσύνη ότι οι όροι που θέσαμε για την ουδετερότητα του άνθρακα μέχρι το 2050 και για την μηδενική ρήπανση, αυτοί οι στόχοι που θέσαμε είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι. Αλλά όχι επειδή βρίσκονται τόσο στο, στα, στα καθήκοντά μου, αλλά γιατί είναι θέμα επιβίωσης του πλανήτη μας και ήδη οι, νέοι μας λένε «Μα τι κάνετε». Θα πρέπει λοιπόν για όλα αυτά να καινοτομήσουμε πολύ περισσότερο και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος που έχουμε σε κάποιες τεχνολογίες. Χαμηλή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, φιλοπεριβαλλοντικά αυτόνομα οχήματα, υδρογόνο, συνδεδεμένα αντικείμενα, υγεία, μικροελεκτρονικά, συσσωρευτές, μπαταρίες είναι συγκεκριμένα θέματα. Κινητικότητα, η διάγνωση, η ορθή ιατρική διάγνωση, πιο φιλοπεριβαλλοντική τρόπη παραγωγής ενέργειας. Επίση, θα πρέπει να υιοθετήσουμε την προσέγγιση τη αξιακή αλυσίδα. δηλαδή όλοι οι βιομήχανοι ενό κλάδου να συνεργάζονται προ την υλοποίηση του κοινού στόχου. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα, γίνουμε, θα μείνουμε εξαρτημένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, θα μπούμε σε μια τεχνολογική υποτέλεια που είναι ανυπόφορη. Για μένα η καλύτερη προστασία είναι η αριστεία. Θα πρέπει να πεδίουμε από κοινού, ε, αξιοποιώντα του καλύτερου εγκεφάλου, ε, του μηχανικού μα τους ε, δημιουργικούς επιστήμονές μας. Το κάναμε για τα ε, διαστημικά προγράμματα, το Γαλιλαίο, το Έγνος, το Κοπέρνικος. Θα πρέπει αυτή τη μέθοδο που απέφερε καρπούς να τα χρησιμοποιήσουμε και στη βιομηχανία. Τα κοινά βιομηχανικά προγράμματα, δηλαδή τα σημαντικά προγράμματα κοινού ε, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, όχι μόνο από τα γραφεία των Βρυξελών, αλλά σε συνεργασία με τη βιομηχανία. Έτσι θα ενισχύσουμε από κοινού την εσωτερική αγορά, την ενιαία αγορά και εντός και εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και τώρα περνάω στα αγγλικά. Όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτή. Κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να προστατευτούμε ε, εγκαταλείποντας ε, το, το άνοιγμα προς τα έξω, αλλά όχι, η Ευρώπη έχει διαμορφωθεί από την ανταλλαγή ε, προϊόντων και ιδεών. Δεν μπορούμε να κλείσουμε απέναντι στον έξω κόσμο. Από την άλλη, θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε να είναι δίκες οι ε, παγκόσμιες ανταλλαγές. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην προστασία και τον προτεξιονισμό. Για να είμαστε ανοιχτοί, αλλά όχι ευάλωτοι, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα εργαλεία μας για την καταπολέμηση του άδικου ανταγωνισμού. Ξέρω ότι ο Φιλ Χόγκαν πρόσφατα σας ε, περιέγραψε τις ιδέες του για το θέμα αυτό, να ε, έχουμε αμοιβαιότητα όσον αφορά τις δημόσιες ε, συμβάσεις και να εξετάσουμε και τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, όσον αφορά τις τεχνολογίες του μέλλοντος, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη ή το 5G, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καθορίσει τους παγκόσμιους κανόνες. Το κάναμε αυτό με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων που στήριξε ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θέλουμε να το ξανακάνουμε. Θα μιλήσω γερμανικά τώρα. Και τέλος η πέμπτη μου προτεραιότητα. Η καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων ε, και η συμμετοχή τους ε, στις μεταβολές αυτές. Όλα αυτά θα τα πετύχουμε μόνο αν ακολουθήσουμε τις αρχές μας. Μαζί με την Μαγκρέτε Βεστάγκερ, τις πρώτες 100 μέρες της εντολής μας θα ε, εργαστούμε πάνω στα θέματα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα φροντίσουμε να έχουμε νέα ε, νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές ε, υπηρεσίες. Αναθεώρηση δηλαδή της νομοθεσίας που εκπονήσαμε πριν 20 χρόνια. Θα ασχοληθούμε με την πλατφόρμα για την προστασία των χρηστών και τη μη διάκριση μειονοτήτων, θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την προστασία των παιδιών. Θα πρέπει να υπερασπίσουμε τις ε, ελευθερίες μας, ε, την ελευθερία του τύπου και την καλλιτεχνική ελευθερία πάνω απ' όλα. Το πώς ε, θα χειριστούμε τις πληροφορίες είναι το σημαντικό, αλλά η σχέση ελευθερίας και ασφάλειας δεν είναι απλή υπόθεση. Σε συνεργασία μαζί σας ε, θα προσπαθήσω να καταλάβω το πρόβλημα καλά προτού αναλάβω οποιαδήποτε δράση. Όσο περισσότερη ψηφιοποίηση έχουμε, τόσο πιο σημαντική είναι η κυβερνοασφάλεια. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά και να δημιουργήσουμε μία μονάδα που να μπορεί να ενεργήσει σε περίπτωση ε, κυβερνοπιθέσεων. Όσο προχωράει όμως η ψηφιοποίηση, τόσο πιο αποφασιστική σημασία είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων. Στόχος μας θα πρέπει ε, να είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκπαίδευση ε, σε ε, θέματα ψηφιοποίησης και ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει σχέδιο για την ψηφιοποίηση. Όταν ήμουν Ευρωβουλευτής, είχα τη δυνατότητα να συμμετέχω, να προεδρεύω στην ομάδα για την ε, καταπολέμηση της φτώχειας. Ε, γνωρίζω ανθρώπους ε, που έχουν γνωρίσει τη φτώχεια. Εάν με υποστηρίξετε ως ε, επίτροπος θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό, προστατεύοντας όλους τους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω, left behind όπως λέμε. Θέλουμε οικονομία κοινωνική και με αλληλεγγύη και μέσα σε πέντε χρόνια θα μετρήσουμε την επιτυχία μας ανάλογα με το κατά πόσο έχουμε προστατεύσει τους ασθενέστερους ε, για να ε, μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ψηφιοποίηση. Περνάω στα γαλλικά. Η κυρίαρχη αυτή η Ευρώπη που θα δείχνει αλληλεγγύη και θα ευημερεί είναι αυτό που θέλουμε. Και ευχαριστώ και την οικογένειά μου για την αγωγή που μου έχει δώσει και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να απευθυνθώ και να θυμηθώ μάλλον τους γονείς μου παρόλο που τους έχω χάσει. Ε, Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τον να έχει κανεί ε, ισχυρή εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκή. Έχω εργαστεί πολλά χρόνια στα ευρωπαϊκά θέματα, κοντά στον Ρωμανό Πρόντι, ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Eurosystem. Έχω κάνει έρευνα, έχω δημοσιεύσει πολλά βιβλία και έχω αναλάβει πολλέ πρωτοβουλίε πολιτών, όπω το Ευρωπαϊκό Κίνημα στη Γαλλία για τέσσερα χρόνια και σε άλλα ε, διεθνή κινήματα. Πολλέ φορέ η δραστηριότητά μου έχει προκαλέσει ερωτηματικά, όμω όλα εντάσσονται σε αυτήν την πορεία μου. Και ε, το Συμβούλιο για το Μέλλον τη Ευρώπη συγκεντρώνει ακαδημαϊκού, πολιτικέ προσωπικότητε, πολλού από αυτού με του οποίου συνεργάστηκα για θέματα όπω η διακυβέρνηση ή η άνοδο των ευρωφοβικών και αντιευρωπαϊκών κινημάτων. Γι' αυτό, κυρίε και κύριοι, ε, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε μια δεκαετία κρίσης οικονομική, κοινωνική ε, και το είδα στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο όταν ενισχύσαμε το οικονομικό πλαίσιο καθώς και την κρίση τη μεταναστευτική που έχει δημιουργήσει μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ Ανατολή και Δύση. Υπάρχουν πολλά πληγέ αυτή τη στιγμή στα σύνορα τη Ευρώπη. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάζουμε προ τα πίσω, αλλά το μέλλον. Πρέπει να συμπαρασύρουμε του Ευρωπαίου για να κάνουμε πράγματα μαζί. Να μην αναρωτιόνται από πού ερχόμαστε, αλλά πού πηγαίνουμε όλοι μαζί. Και θέλω να συνεργαστώ με όλου σα και με του συναδέλφου μου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ΕΟΚΕ, με την ε, Επιτροπή των Περιφερειών, με όλε τι δυνάμει, τι ε, ζωτικέ δυνάμει τη κοινωνία, τη οργανώση των πολιτών και ω πρώην Ευρωβουλευτή. Κυρία Πρόεδρε, και υπάρχουν εδώ συντονιστέ τη Επιτροπή ΕΚΟΝ Θέλω πραγματικά να έχουμε μια στενή συνεργασία, διαρκή συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναλαμβάνει τι πρωτοβουλίε και του Ευρωκοινοβουλίου που είναι ουσιαστικά το άλλο σκέλο τη νομοθετική διαδικασία. Θέλω σε κάθε ε, φάση της νομοθετικής διαδικασίας, σε κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε, να μπορούμε να ε, έχουμε συνομιλίες. Δεν ξέρω αν θα συμφωνεί μαζί μου ακριβώ όλο το υπόλοιπο το κολέγιο των Επιτρόπων, αλλά θέλουμε με αμοιβαίο σεβασμό και συνομιλίε επικοινωνία να εξασφαλίσουμε μια καλή συνεργασία και για το μέλλον. Σα ευχαριστούμε στη διάθεσή σα, κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρ για την προφορική σα δήλωση. Περνάμε τώρα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων που θα θέσουν τι ερωτήσει. Ο πρώτο είναι ο κύριο Φρανσουά Ζαβιέ Μπελαμή εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Καλημέρα σας. Για να αντιμετωπίσουμε ε, τις προκλήσεις βιομηχανίας, του εμπορίου και της άμυνας, θέλουμε μια ισχυρή βιομηχανία, αλλά και την απαραίτητη εμπιστοσύνη δράσης. Ως Υπουργό Άμυνα στη Γαλλία προτιμήσατε να παρατηθείτε για μια δικαστική έρευνα που γινόταν για την εντολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είπατε ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της δημόσιας δράσης και αυτό υπερέχει του προσωπικού συμφέροντος και η τιμή ε, των υπουργών δεν θα πρέπει να διακυβεύεται σε πολεμικές από τις διάφορες ε, πλευρές. Είπατε ότι πιστεύετε τα κράτα στην Ευρώπη και μιλήσετε για διάφορες απαιτήσει. Ε, βέβαια, πρόσφατα αναγκαστήκατε να επιστρέψετε ένα διόλο μελιτό ποσό και συνεχίζεται και η δικαστική έρευνα. Βέβαια, δεν είμαστε εδώ για να σας κρίνουμε για να σας δικάσουμε, αλλά με τους συναδέλφους του ΕΛΚ θα ήθελα να σας ε, θυμίσουμε τα λεγόμενα σας πώς να, ε, ε, πώς να πιστέψουμε ότι αυτό που σας απομάκρυνε από τη γαλλική κυβέρνηση θα σας επιτρέψει με την υφαλιότητα και την ανεξαρτησία να υλοποιήσετε τα καθήκοντά σας ως επιτρόπου. Δεν θα πρέπει να εφαρμόσετε τους ίδιους κανόνες εδώ με την εθνική σας πολιτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκουλάρ, χαίρομαι που μου θέτετε αυτή, την ερώτηση, γιατί θα έχω την ευκαιρία να σα απαντήσω. Καταρχήν, το τεκμήριο αθεο... αθωότητας είναι θεμελιώδη ελευθερία και κατοχυρώνεται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, στα οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου και στο γαλλικό σύνταγμα. Για όσου όμω δεν είναι Γάλλοι, θα ήθελα να πω ότι από τη ε, δεκαετία του 90 υπάρχει το θυμικό δίκαιο από τη στιγμή που ένας υπουργό ε, είναι αντικείμενο δικαστικής έρευνας, οφείλει να παραιτηθεί. Ε, το 2017 ξεκίνησε μια δικαστική έρευνα σχέση με την αμοιβή ενό ε, ε, βοηθού της ομάδας μου και τελικά δεν χρειάστηκε να τεθώ υπό έρευνα αλλά έκρινα για λόγους ευθυξίας ε, και λόγω της επιτακτικής ανάγκης ε, που υπήρχε για, ε, για το στρατό στη Γαλλία, την στρατιωτική μας επιχείρηση στο Μαλί αλλά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις, έκρινα, ε, ακούγοντας τη συνείδησή μου, ότι δεν μπορώ να θέσω σε κίνδυνο τη, τα γαλλικά στρατεύματα και τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν εκεί. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Καταρχήν, έδωσα τη μαρτυρία μου στην γαλλική δικαιοσύνη και τελικά δεν συνεχίστηκε η έρευνα. Από ό,τι ξέρω, στα ευρωπαϊκά ζητήματα δεν ισχύει αντίστοιχο έθιμο, αντίστοιχη συνήθεια παρέτησης. Θα ήθελα μόνο να σας πω το εξής. Μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή η αρχή τη ακαιρεότητα και μάλιστα πήρα μία απόσταση από τα πράγματα και τίποτα δεν παραδέχτηκα κύριε Μπελαμή. Δεν ε, ομολόγησα καμία υπετιότητα. Μάλιστα έγινε ευρυθής έρευνα, ε, διαπιστώθηκε ότι ο βοηθός μου εργάστηκε μία με πενταετία και έπρεπε να γίνει κάποια επιστροφή, όχι γιατί εγώ έλαβα τα χρήματα αυτά, αλλά επειδή υπήρξαν προβλήματα τη στιγμή τη παρέτησή του. Έγινε μία αντιπαράθεση εδώ του γαλλικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Και θα ήθελα να σας θερμοπαρακαλέσω όλου να σεβαστείτε το τεκμήριο τη αθωότητας. Κύριε Μπελαμή, έχετε περώτηση. Ευχαριστώ για την απάντηση σα. Το τεκμήριο αθωότητας φυσικά είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα και σε καμία περίπτωση δεν το αφισβητώ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό που υπογραμμίσατε τελευταία στιγμή. Ο κίνδυνος ε, που δημιουργήσετε για το Προεδρείο σας όσο ε, ήσασταν εμπλεκόμενοι σε μια δικαστική έρευνα. Καμία στιγμή ε, της παρέτηση σας δεν είπατε, ούτε την δεν μιλήσατε ούτε για τη δημοκρατία, την προοπτική της δικαστικής έρευνας, ούτε για αυτό το εθνικό δίκαιο τη γαλλική διοίκηση. Ενώ είπατε ότι θα τηρήσετε τις ε, ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είστε προσιλωμένοι στην ευρωπαϊκή ιδέα που κανονικά θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά από αυτά που ισχύουν στη, στη γαλλική ε, ενόμη τάξη. Θέλουμε μια ισχυρή στρατηγική στον τομέα σας για να ανακτήσουμε την ε, ζωτικότητά μας, την βιομηχανική και την οικουμενική. Κάτι λοιπόν που θα ήταν και επικίνδυνο για το Γαλλικό Υπουργείο και ενώ συνεχίζεται, είναι εκρεμή έρευνα στην ΟΛΑΦ, άσχετα από την υπετιότητά σας, φυσικά δεν μπορώ να προδικάσω τη μία ή την άλλη ε, κατηγορία, αλλά πώς είστε σίγουροι ότι αυτή η εκκρεμούσα δικαστική έρευνα δεν θα επηρεάσει την υφαλαιότητα και την αμεροληψία σας κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων σας. Ε, νιώθω ε, πολύ γαλήνια και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν είμαι δεν με έχουν υποβάλει σε έρευνα. Βέβαια, η Όλαφ ε, αυτόματα επιλαμβάνεται όταν ξεκινά μια διαδικασία σε μια χώρα, οπότε περιμένω την δικαστική απόφαση, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έκρινε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα σύγκρουσης συμφερόντων, γι' αυτό επέτρεψε τη διοργάνωση ακρόασης, κάτι που συνιστά ένα καινούριο στοιχείο της διαδικασίας. Απλώς το λαμβάνω υπόψη και νιώθω πολύ άνετα όχι ότι περιφρονώ τη, τα ευρωπαϊκά αξιώματα και το δείχνει και η σταδιοδρομία μου, αλλά νομίζω το θέμα τα, της εμπλοκής ανθρώπινης ζωής είναι τελείως διαφορετικής φύσης. Επίσης υπάρχουν κάποια άρθρα που γράφονται στον τύπο, αλλά τι, τι ξέρετε σε από αυτά που είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για το εθνικό δίκαιο που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις στη Γαλλία. Με, τις, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Άκουσε τη συνείδησή μου και έλαβε την απόφαση τότε ω Υπουργό ε, Άμυνα και τώρα με απόλυτη συνείδηση έρχομαι εδώ ενώπιον σα και ζητώ την εμπιστοσύνη σα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σχάλτεμο ε, από το SND. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλώ ορίσατε πάλι στο κοινοβούλιο, κυρία Κούλαρ. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να συνεχίσω προ την ίδια κατεύθυνση. Πριν πέντε χρόνια στι ακροάσει ήσασταν στη δική μα θέση και είπατε για τον ε, συμπατριώτη σας Μοσκοβισή ότι πιστεύετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ε, την ε, συμπεριφορά ή την προσωπικότητα κάποιου. Δεν πιστεύετε ότι μπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο για σας. Έχετε μία υπόθεση του Όλαφ, έχετε πληρώσει, έχετε επιστρέψει 45.000 ευρώ. Το είχατε τονίσει εσείς για το Μοσκοβισή πριν τόσα χρόνια. Τώρα πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα σέβομαι απολύτως την δουλειά που κάνετε και την έχω κάνει και η ίδια και ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός αυτής της ακρόασης. Να υποβληθώ σε όλες τις ερωτήσεις. Όταν πέρασα από ακρόαση ο κ. Μοσκόβηση και δεν ε, θα ήθελα να τον ανακατέψω περαιτέρω σήμερα, είναι ε, το θέμα ήταν ότι τότε η Επιτροπή είχε να κάνει με το πώ τα κρατικά δημοσιονομικά ε, αποτελούσαν αντικείμενα διαχείριση και χωρί να υπάρχει και προσωπική ανάμεξη. Αυτή τη στιγμή είναι άλλο το πολιτικό στοίχημα. Τότε υπήρχε η κρίση της Ευρωζώνης, υπήρχε έλλειψη εμπιστοσύνης. Κάποια κράτη-μέλη σέβονταν λιγότερο το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τελείως διαφορετικές συνθήκες. Για το θέμα των ποσών που ε, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το θεσμικό σας όργανο ε, και ο Γενικός Γραμματέας διοργάνωσε μια δεξιοδική έρευνα διοικητικού χαρακτήρα για να δει αν ο τοπικός βοηθός που εργαζόταν για μένα εργάστηκε πραγματικά ή όχι. Και πάντα ήταν ναι, για μια πενταετία. Αυτό που αμφισβητήθηκε ήταν και αυτό συμβαίνει συχνά σε ε, εργοδότε. Ξέρω ότι πολλοί ε, σε μικρομεσαίε στη Γαλλία, αν μα ακούνε, θα, το, θα θυμηθούν του εαυτού του. Έχουν κάποιοι έναν εργαζόμενο, ένα μισθωτό, που θέλει να διακόψει τη σύμβαση του εργοδότη, αλλά δεν θέλει να τον τιμωρήσει, να του δημιουργήσει προβλήματα και να τον απολύσει. Οπότε ξέρει ότι θα έχει δυσκολίε να βρει άλλη θέση. Και περνάνε εβδομάδε. Ε, πήρε λίγο καιρό για να διακοπεί η σύμβαση. Ήταν θέμα διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Εάν κοιτάξετε τι αποφάσισε σε Γενική Γραμματεία, το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του οργάνου σα, θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου δικαστική υπόθεση. Είναι μια διοικητική επαλήθευση και είναι θέμα διοίκηση. Είναι θέμα διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Δεν ήταν καθόλου ποσά τα οποία έλαβα, κυρία Σαλντεμόζε, να είστε βεβαία. Ε, ρωτήστε του συνεργάτε σα. Ε, σε περίπτωση απόλυσης θα πήγαινε στο δικαστήριο υπεύθυνη εγώ ίδια. Όμως ε, υπάρχει μια δυσκολία στο Κοινοβούλιο με τον τρόπο που έχει συνταχθεί το εσωτερικό κανονισμό ό,τι αφορά το καθεστώ των βοηθών. Σας ευχαριστώ. Η ε, δευτερολογία της κυρίας Σάλτεμόζε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην επιστολή ανάθεση καθηκόντων τονίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τη συμπεριφορά ή την ακυρεότητά σα. Εγώ νομίζω ότι 45.000 ευρώ είναι πολλά χρήματα, γι' αυτό έθεσα την ερώτηση. Ε, για μένα δεν ετέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Ήθελα λοιπόν να το ε, ρωτήσω αυτό. Δεν πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ε, καθαροί οι υποψήφοι επίτροποι και να ε, έχουν ε, αδιαφυσβήτητη ακαιρεότητα. Είμαι πεντακάθαρη. Έχω σεβαστεί όλη τη διαδικασία και του κανόνε που έθεσε το γραφείο του Γενικού Γραμματέα. Σέβομαι την απόφαση του Γενικού Γραμματέα και του Κοινοβουλίου. Το πόσο σε τι αναλογεί. Σε μισθού και σε κοινωνικέ εισφορέ σε ασφορές, σε ταμεία. Δεν θα ήθελα να περάσουμε σε συζήτηση επί των λεπτομεριών, αλλά είμαι βεβαίω, αν το κοιτάξετε, και χαίρομαι που είμαι στο ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη χρηματοδοτούν την κοινωνική ασφάλεια, ε, την κοινωνική πρόνοια και εδώ και αλλού. Υπευλήθη λοιπόν στην ε, απόφαση του Γενικού Γραμματέα ε, του Ευρωκοινοβουλίου που εφάρμοσε μια νομολογία πολύ αυστηρή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι όταν ε, κάποιος βοηθός εργάζεται για σας μπορεί να λάβει κατά τους καταβληθέντα. Ρωτήστε το γραφείο του ε, Γενικού Γραμματέα. Δεν είναι καταδίκη και δεν υπήρξε τιμωρία. Δεν πληρώθηκαν για αυτά, τα χρήματα. Ευχαριστούμε κυρία Χαράντσοβα από την Renew. Thank you very... Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητή Σίλβη, όπως και πολλοί άλλοι εδώ σε γνωρίζω καλά, γνωρίζω πόσο σκληρά εργάζεσαι, ξέρω πόσο προσιλωμένη είσαι στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και είμαι πεπισμένη, γνωρίζω ότι έχεις τις, τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση αυτή και ε, θα κάνεις καλά τη δουλειά σου. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω σήμερα είναι, έχεις το θάρρος, την τόλμη να υπερασπιστείς την εσωτερική αγορά και τις ελευθερίες που παρέχει η εσωτερική αγορά. Στην επιστολή ε, ε, ανάθεσης καθηκόντων αναφέρεσαι στην ψηφιοποίηση ως ένα από τα βασικά σου ε, καθήκοντα ή τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ε, συμφωνώ ότι χωρίς ε, υπηρεσίες η εσωτερική αγορά δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη. Είχαμε τον κύριο Βόλκενστάν και τον κύριο Μπαρνιέ που υπερασπίστηκαν την εσωτερική αγορά και οι δύο την υπερασπίστηκαν, καταπολέμησαν ε, τα διάφορα συμφέροντα και στην πατρίδα τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ λοιπόν, έχεις την τόλμη να συνεχίσεις το έργο αυτό και θα μπορέσεις να διευρύνεις την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρ. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ που θυμηθήκατε τη δουλειά μου. Νομίζω ότι όσοι βρίσκονταν εδώ στο Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι έχω δώσει αρκετού αγώνε για την ισότητα ανδρών γυναικών, για την Τραπεζική Ένωση, για την ε, αναθεώρηση του ε, Συμφώνου Σταθερότητα. αλλά δεν έχω την ελαζονία να πιστεύω ότι μόνο ε, ο επίτροπο έχει το μονοπόλιο τη τόλμη. Δεν είναι έτσι, γιατί στο λόγο μου, στην ομιλία μου αναφέρθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει κατά κάτι μέλη να συμφωνούν. Πρέπει όλε οι επιχειρήσει, ο της βιομηχανία, όλοι ο χώρο τη οικονομία, να είναι πεπισμένοι ότι η Ευρώπη αποτελεί ατού, αποτελεί πλεονέκτημα. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν και συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Σαφώ υπάρχει δυναμικό ανάπτυξη, ε, υπάρχουν θέσει απασχόληση που συνδέονται απευθεία με τις βελτιώσεις που θα επιφέρουμε στα κείμενα περί υπηρεσιών. Έχω εμπειρία από αυτό το χώρο, αλλά το έχω πει και στο παρελθόν. Έχουν γίνει πολλέ προσπάθειε προηγουμένω που κατέληξαν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα μέρο του πληθυσμού να το βάλουμε στο περιθώριο με άγχη τα οποία τα καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνω το κλίμα στο οποίο αναφέρεστε. Όμω, εμεί θα πιάσουμε κατευθείαν μια πράξη για την νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Θα κοιτάξουμε τη συνεργατική οικονομία. Θα κοιτάξουμε να υπάρχει περισσότερο enforcement, περισσότερη επιβολή των, ε, και εφαρμογή των κανόνων και θα δούμε του τομεί ε, ξεχωριστά αυτού με του οποίου θα ασχοληθούμε. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα κατευθείαν, βέβαια. Και το σημαντικό είναι να συνεργαστούμε και μαζί να καταφέρουμε να συμπαρασύρουμε του πολίτε. Ε, για τι χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορέ σε σχέση με μια χώρα όπω η Γαλλία που έρχομαι εγώ. Ε, έχουν διαφορετικέ παραδόσει, διαφορετικέ αξίε, δεν είναι ακριβώ ταυτόσιμε. σω να μην έχουμε ακριβώ τι ίδιε προτεραιότητε λοιπόν. Γι' αυτό πρέπει συνεχώ να συνομιλούμε και να επικοινωνούμε και θα κάνω ό,τι μπορώ με όλε μου τι δυνάμει, με όλη μου την ενέργεια για να προχωρήσει όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Σα ευχαριστούμε. Ε, περώτηση. Όσον αφορά την πράξη για τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Υπάρχουν διάφορε ιδέε για το πώ να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Ε, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή τη σχετική συζήτηση. Είμαι βέβαιη ότι και το Κοινοβούλιο θα έχει λέγει στην υπόθεση αυτή. Η ερώτησή μου όμω είναι, σκοπεύετε με την πράξη αυτή να ενισχύσετε την ελεύθερη ε, κυκλοφορία των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Μπορείτε να μου υποσχεθείτε, να δεσμευτείτε ότι δεν θα δημιουργήσετε νέα εμπόδια εντό Ευρώπη. Η κυρία Γκουλάρ. Γι' αυτό προασπιστήκαμε από κοινού την αγορά κατά τι διαπραγματεύσει για τον Brexit. Είναι τέσσερι θεμελιώδεις ελευθερίες και επιμένω. Ε, Ίσως αυτό θα πρέπει και να υπογραμμίσουμε και στους πολίτες, να το προβάλλουμε για να δουν τα ωφέλη, για να το αντιληφθούν. Ναι, ε, είναι οι τέσσερις αυτές ελευθερίες. Η ελευθερία της κυκλοφορίας, η ελευθερία του να εργαστεί κανεί αλλού, να πάει να σπουδάσει, να εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, να μπορεί να πουλήσει προϊόντα. Είναι ελευθερίες. Ε, και η ελευθερία στο διαδίκτυο. Αν δεν κοιτάξουμε να διοργανωθούμε μεταξύ μας, μπορεί να εξαφανιστεί από πολύ ισχυρού φορεί από το διεθνέ προσκήνιο που μπορεί να έχουν την δυνατότητα να διεισδύσουν και να επηρεάσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι λοιπόν η πώληση των υπηρεσιών, είναι η ε, ο δυναμικό χαρακτήρα των νεοφυών επιχειρήσεων, των startup. Γιατί πολλέ φορέ είναι μικρομεσαίε επιχειρήσει και νέοι που εργάζονται. Και επίση πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό ε, στου κανόνε και την νομοθεσία. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε εισάγει ε, κανόνε και φραγμού. Πρέπει απλώ να πείσουμε του άλλου διεθνεί φορεί ότι Πρέπει να πάμε όλοι μαζί στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια. Ε, ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Μαρσέλ Κολάγια από του Πράσινου. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ υποψήφια επίτροπε. Παρά τους 250.000 μόνο στη Γερμανία που διαδηλώνουν και υπογράφουν αναφορές κατά της ε, ε, ευθύνης των παραχών υπηρεσιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να κάνει πιο αυστηρές ε, τις διατάξεις για την ε, ευθύνη αυτή στη νέα οδηγία για τις ε, ψηφιακές υπηρεσίες. Και παρόλα αυτά στη Γαλλία έχετε νομοθετικές διατάξεις ε, για ρητορική μίσους που επικρίνεται από μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα online. Η ε, θέση σας, η ε, εθνική και η ρυθμή στη Γαλλία θα επηράσει την, τα καθήκοντά σας ως επιτρόπου παραβιάζοντας την ελευθερία στο διαδίκτυο. Το θέμα της ευθύνης για ρητορική μίσους και παραπληροφόρηση online. Ναι, όμως μερικές φορές δεν θα ήταν πιο επικοδομητικό να επικεντρωθούμε στην εξέταση της ακρίβειας των στοιχείων και στη διαφήμιση για να λύσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα, γιατί αφορά την ελευθερία η Ευρώπη είναι η μόνη παγκόσμια οικονομία και η μόνη κοινωνία που έχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που εξασφαλίζει και εγγυάται την ουδετερότητα του διαδικτύου. Και αυτό δεν αφισβητείται από το νέο σχέδιο οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η επικαιροποίηση που γίνεται με το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό φορέα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες φροντίζει για την σωστή εφαρμογή αυτής της αρχής. Βέβαια, έχουμε εδώ, πριν από, εδώ και 20 χρόνια την ιδέα της ε, ε, περιορισμένης ευθύνης. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, 20 χρόνια είναι τεράστια χρονική διάρκεια. Δεν αφισβητούμε την αρχή του liability της ευθύνη, δεν κάνουμε ρήξη και έλεθες αλλαγές, αλλά απλώ επιτρέπουμε και είναι προσυζήτηση το θέμα. Είναι μια διαδικασία που θα κάνουμε από κοινού, να εξετάσουμε σχολαστικά πού θα εφαρμόζεται αυτή η ευθύνη. Αναφερθήκατε στο θέματα της ρητορικής μίσους, ε, της υποδάβλησης του μίσους μέσω του διαδικτύου. Εγώ δεν είμαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιβάλλω τη γαλλική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι αυτό το σκεπτικό μου, ούτε η πρόθεσή μου. Θα πρέπει όμω να κοιτάξουμε κατάματα ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Έχουμε στο διαδίκτυο και κάποιου που ε, καλλιεργούν το μίσο, υποδαβλίζουν το μίσο, στιγματίζουν κάποιε κοινότητε για τη θρησκεία του και κάνουν διακρίσει ε, ή ε, παροτρύνουν σε διακρίσει και μίσο με σημαντικέ συνέπειε. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ τη ελευθερία τη έκφραση και αυτή τη συμπεριφορά. Και η επιλογή πολιτική που θα γίνει είναι επιλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά έχουμε και το Συμβούλιο, που επίση εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώ θα προτείνει το κείμενο, εσεί θα το τροποποιήσετε. Και έρχομαι μπροστά σα χωρίς καμία υπεροψία και αλαζονία, γιατί δεν έχω έτοιμη λύση. Τη λύση θα τη διαμορφώσουμε από κοινού, αν συνεργαστούμε. Επερώτηση, συγγνώμη, κύριε Κολάγια, συμπληρωματική ερώτηση. Έχω επερώτηση για τα θέματα που αναφέρατε στην αρχή. Είναι σημαντικό για την ομάδα μας γιατί ο γαλλικός τύπος είπε ότι όσο ήσασταν ευρωβουλευτής, ε, λαμβάνατε 10.000 ευρώ το μήνα για 27 μήνες μεταξύ του 2013 και 2014 από το ε, Ινστιτούτο Μπέργκρουεν, φιλοευρωπαϊκό. Και είπα και αναφέρθηκε ότι ήσταν σύμβουλο Ευρωπαϊκή Πολιτική στο Ινστιτούτο αυτό. Είχατε στενέ επαφέ με, την, τον διευθυντή του Ινστιτούτου. Βέβαια αναφέρεται ότι είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση αυτό το Ινστιτούτο και δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων τότε με την εντολή σα τη βουλευτική σα εντολή. Το βουλευτικό όμω έργο είναι μια πλήρη απασχόληση. Πώ συνδυάσετε τη βουλευτική σας έδρα με, τη παροχές, με τις παροχές συμβουλών σε αυτό το Ινστιτούτο. Ήταν άσχετη η επερώτηση σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, ενώ κανονικά θα πρέπει να συνδέονται. Είστε ελεύθεροι να απαντήσετε ή να μην απαντήσετε. Φυσικά και θα απαντήσω γιατί είμαι υπέρ τη ελευθερία και στο διαδίκτυο και γενικώ. Από μόνιμα ανέφερα αυτή τη συνεργασία με το Think Tank, το Ινστιτούτο Berggren, ήταν ένα φιλοευρωπαϊκό think tank, συνεργάστηκε κυρίως με Ευρωπαίους στα πλαίσια αυτού του Ινστιτούτου. Όλα τα είχα δηλώσει, όλα ήταν διαφανή και νόμιμα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεπε, τουλάχιστον όσο εγώ δούλευα, ε, την παράλληλη άσκηση επαγγελματική δραστηριότητα. Τώρα, αν αυτό είναι σημαντικό ή όχι, είναι θέμα προσωπική επιλογή του Ευρωβουλευτού. Υπήρχε δυνατότητα και σε ένα κράτο δικαίου μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, γι' αυτό και σα απαντάω. Δεν μπορούμε όμως να ρίχνουμε υπόνοιες για κάποιον επειδή δούλευε. Δούλευε γιατί. Δούλευε για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και μάλιστα ε, το Μάιο του 2013 συνάντησε εκπροσώπους του Ινστιτούτο Μπέργκρουεν σε μια διάσκεψη του, του Πανεπιστημίου Πολιτικών Επιστημών για την απασχόληση των νέων. Σε μια τέτοια διάλεξη λοιπόν, γιατί ούτως ή άλλως ε, ε, και οι υπουργοί από τι χώρες Ευρώπη Ευρώπης ε, συζητούν για το θέμα της απασχόληση των, των νέων. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξε τους ίδιους στόχους και φιλοδοξίες μέσω όμως μιας άλλης ιδιόδου του Ινστιτούτου αυτού. Κύριε Γιωρό, από την ομάδα Ταυτότητα Δημοκρατία. Ε, κυρία μου, εδώ Παρατηθήκα από την κυβέρνηση Μακρόν ε, για τι έρευνε που αφορούσαν την κοινοβουλευτική σα δραστηριότητα. Δέχω την επιστολή του Όλαφ που ε, λέει ότι είστε μόνοι υποψήφιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είστε ε, ε καθεστώ έρευνα. Δεν είστε άξια να είστε μέλο τη γαλλική κυβέρνηση, αλλά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Βρυξέλλη. Ποιο κερδίζει 13.000 ευρώ το μήνα για να κάνει τηλεφωνήματα, κυρία μου. Θα είχατε χρηματοδοτήσει με αυτό το ποσό ό,τι θέλατε όσο ήσασταν Ευρωβουλευτή. Έχετε γράψει κάτι διαφορετικό από αυτό το σημείωμα 13 σελίδων για τα 13.000 ευρώ επί τρία χρόνια. Ναι, γράψετε μια έκθεση. συντάξετε μια έκθεση στην περασμένη σα θητεία για τη δημιουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αυτή η διεθνιστική θεώρηση υπέρ τη παγκοσμιοποίηση μα ανησυχεί. Θέλουμε να σεβαστούμε τι ταυτότητε και την εθνική κυριαρχία των ευρωπαϊκών κρατών. Τι υπηρεσίε προσφέρατε ε, στους πολίτες με τέτοιε αμοιβέ. κυρία μου, και με αυτά που κερδίσατε, καθώ και με την αμοιβή σα από το Ινστιτούτο Μπέργκμαν που ξεπέρασε τα 300.000 δολάρια. Κυρία Βουλευτά, ε, έχω Νομίζω ήδη απαντήσει, αλλά θα τα επαναλάβω. Δεν μπορεί κανείς να αμαυρώνει την εικόνα κάποιων χωρίς να προσφέρει αποδείξεις. Δούλεψα για ένα think tank με ενέργειες που είχαν να κάνουν με διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, με μελέτες. Συνεργάστηκα με πολλούς και οι συνεργάτες μου το επιβεβαιώνουν. Οι στόχοι ίσως να μην σας άρεσαν, αλλά έχετε κάθε δικαίωμα γιατί είμαστε σε καθεστώς δημοκρατίας. Ε, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια κυβέρνηση πιο παγκοσμιοποιημένη. Εσείς μπορείτε να μην συμμετέχετε σε αυτό το όραμα. Όμως το 2013 βρισκόμασταν σε μια φάση πραγματικά ιδιαίτερα οξία της ε, κρίσης. Και νομίζω ότι ο σκοπό εδώ αγιάζει τα μέσα. Ό,τι τρόπο είχαμε για να προσελκύσουμε του πολίτε ή να του βοηθήσουμε ήταν καλά. <clears throat> για την ανεργία λοιπόν ε, κάποιοι μου είπαν να μην συζητάω με άλλου που έχουν διαφορετικέ απόψει. Εγώ θεώρησα ότι ήταν πολύ σημαντικό να έρθω σε επαφή με, πολλούς, ε, με πολλέ ισχυρέ προσωπικότητε. Με ανθρώπου όπω ο Μόντι, ο Φερχόφστα, τον Γκονσάλε, ε, ο, Άντωνι Γκίντεν, πρώην πολιτικού αρχηγού, διανοωμένου, για να προχωρήσει το όλο θέμα. Τώρα, ότι είχα φανταστεί ότι θα δημιουργούνται κάποια μέρα προβλήματα, σε καμία περίπτωση τα, το καταλαβαίνω ότι σας φαίνονται υψηλά τα ποσά. Παχυλέ, παχυλή μισθή. Όμως έτσι είναι οι αμοιβέ, οι απολαυέ όσων προσφέρουν ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες διεθνώς. Μπορώ να εργαστώ σε τέσσερι γλώσσε και να διοργανώσω πολύ μεγάλε εκδηλώσει με συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων. Τώρα, ε, ε, αν δεν προστατεύσουμε την ελευθερία του επιχειρήν, θα πρέπει να σκεφτούμε το ίδιο και το τεκμήριο της αθότητας, κυρία μου. Επερώτηση. Ευχαριστώ. Πραγματικά, η είπα, ένα ιστορικό μα τέρο για το καθένα από τα ευρωπαϊκά μα κρατή. Δεν είναι όμω Ευρωπαίοι. Επίση, στο Αμερικανικό Ινστιτούτο αυτό φαίνεται να υπήρχαν διάθεση παρεμβατισμού ε, και όχι ακριβώ μόνο σύγκρουση συμφερόντων. Άρα, άρα φαίνεται με αυτή τη δραστηριότητα να ανακατεύεται διαφορετικά πράγματα και να είναι αρκετά θολή η πραγματικότητα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πανικός. Μόλις σήμερα το πρωί λάβαμε μία επιστολή υποστήριξη από αυτό το λόμπι ε, υπέρ τη αποψηφιότητά σα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια για την οικονομική πραγματικότητα, γιατί η Υποτροπή ε, Νομικών Υποθέσεων αρνήθηκε να μελετήσει τις απολαβές που προήλθαν από αυτό το Think Tank και να μην ξεχνάμε ότι το αφεντικό του Think Tank είχε διασυνδέσεις με τον κύριο Μακρόν. Αυτέ ε, οι προσωπικότητε που λέγαμε ότι θέλουμε να είναι άμεμπτε ω επίτροποι δεν ε, είναι αυτό που εκπροσωπείτε εσεί. Νομίζω ότι τον οδικό σα χάρτη, ε, εάν τον έχετε λάβει από την Καλιφόρνια, δεν θα μπορούσα να σα στηρίξω στην υποψηφιότητά σα ως Ευρωπαίος Επιτρόπου. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά. Παρά, να πω την αλήθεια, δεν περίμενα και την υποστήριξή σα. Αλλά για να πω την αλήθεια επίση και τα γεγονότα να δούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, το είπατε και έχει σχέση με τη ΣΥΠΑ. Είναι ε, ένα φορέα δεν είναι το Πεντάγωνο, δεν είναι η κυβέρνηση, τον είπα. Είναι μέλη τη κοινωνία των πολιτών με του οποίου συζητάμε. Ε, πρέπει να υπάρχει κάποια διάκριση εδώ, κάποιο διαχωρισμό μεταξύ των κυβερνώντων και των ιδιωτών. Ο κ. Μπερνγκό δεν είναι, είναι είναι Γερμανό και ίσω αυτό να μην σα αρέσει. Ε, είναι Ευρωπαίο. Μεγάλωσε στο Παρίσι, καταγόμενο από την Γερμανία και τώρα είναι στη ΣΥΠΑ. Οι διατλαντικέ σχέσει ε, ω πραγματικότητα είναι πολύ σημαντικέ για πολλά θέματα που μα απασχολούν. Έχω συνεργαστεί με Αμερικανού, ε, σεβόμενοι την ανεξαρτησία του και εκείνη τη δική μου. Δεν βλέπω γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι, ε, ε να είναι μεμπτό, αξιόμεμπτο. η Καλιφόρνια είναι το λίκνο πολλών ε, μεγάλων επιχειρήσεων που είναι σημαντικέ για τη διεθνή οικονομία. Και πραγματικά εγώ χαίρομαι που είχα αυτή την εμπειρία την επαγγελματική. Μάλιστα. Επόμενο ομιλητή είναι ο Άνταμ Μπιέλαν. Εκπροσωπεί το, την ομάδα μεταρρυθμιστών συντηρητικών. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Οριστήσα Επίτροπε, ιδιωτικά και δημόσια εργαστήρια έρευνας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο υπόλοιπο κόσμο ασχολούνται με ε, την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς μέσα στις πρώτες 100 μέρες θέλετε νομοθεσία για αυτές τις τεχνολογίες που τώρα αναπτύσσονται. Πόσες μέρες θα χρειαστείτε για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας περί υπηρεσιών. Συμφωνώ με τη γραπτή σας απάντηση ότι ε, η πιο ολοκληρωμένη αγορά υπηρεσιών θα βοηθήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεραιότητες σας αντικατοπτρίζουν την αρχή αυτή. Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ευρύτατος κλάδος απέραντος ε, το προσεγγίζω με ταπεινοφροσύνη, γιατί κάποια πράγματα θα τα κάνουμε μέσα στις 8 μέρε. Ανέλαβα την ε, ευθύνη και η εκλεγμένη πρόεδρο και η εκτελεστική αντιπρόεδρο Φεστάγκερ με πυγμή και αποφασιστικότητα και θα στηριχθούμε στο έργο των προκατόχων μα και θα σκεφτούμε και το δεοντολογικό ζήτημα κατά τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και θα στηριχθούμε σε όλα αυτά. Όπω είπα όμω και πριν από λίγο για τι υπηρεσίε ή για το θέμα της ευθύνης στο διαδίκτυο, είναι ένα τέτοιο απέραντο ζήτημα που θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε. Έχουμε φυσικά κάποιες αρχές που θα ε, μας καθοδηγήσουν, αλλά φυσικά το αποτέλεσμα των εργασιών θα πρέπει να γίνει μετά από συνεργασία μεταξύ μας. Και θα ήθελα να πω και στους πολίτες κυρίως που μας ακούν ότι δεν πρόκειται για μια αφηρημένη συζήτηση. Μιλούμε για τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στους ε, γιατρούς να κάνουν ακριβέστερη διάγνωση. Πρόκειται για τεχνολογίες που θα ε, κάνουν εξακρίβωση πληρωμών. Αυτό είναι χρήσιμο για τις τράπεζες. Επίσης, ε, είναι τεχνολογίες προηγμένες, αλλά θα πρέπει να τις φοβόμαστε. Απλώς θα πρέπει να τις πλαισιώσουμε προσεκτικά, γιατί η χρήση, μαζική χρήση αλγορίθμων σε μεγάλη κλίμακα ίσως δημιουργήσει διακρίσεις. Ίσως, αν το προφίλ σας δεν εμπίπτει σε κατάλληλα πλαίσια, σας οδηγήσει σε μια απόρριψη χορήγηση δανείου από όλες τις τράπεζες. Θα κάνουμε λοιπόν σε έφθετο χρόνο πρόταση που φυσικά θα τη λάβετε και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν χωρίς να ξεχνούμε και τον παραδοσιακό βιομηχανικό κλάδο που επίσης θα πρέπει να περάσει στη νέα εποχή. Και η προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται από το πρίσμα της προσφοράς της τεχνητής νοημοσύνης στους πιο παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας. Έχετε περώτηση κύριε Μπιέλαν. Ε, ο προηγούμενος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς ε, ε, δυσκολεύτηκε να πείσει τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του. Επίσης, διαπίστωσε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές μπορεί να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια της ε, νομοθετικής διαδικασίας. Ε, σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να αποσύρετε τις ε, προτάσεις προτού γίνει ζημιά. Καταρχήν θα ήθελα να πατήσω φόρο τιμή στο έργο της προκατόχου μου, της κυρίας Μπιανκόφσκα. Και δεν αρκεί η τόλμη σε έναν επίτροπο και το θάρρος έχουμε μια γενική κινητικότητα και μια κινητοποίηση μάλλον και από πλευράς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, μια έκκληση για να προχωρήσουμε και με όσα συμβαίνουν με το Ηνωμένο Βασίλειο που μας έδωσε μια λυπηρή απόδειξη αλλά ότι η ενιαία αγορά έχει αξία θα πρέπει πιστεύω πρώτα απ' όλα ε, κύριε Ευρωβουλευτά, να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στα ζητήματα που μας διχάζουν. Δεν είναι αυτά τα πιο σημαντικά. Το πιο σημαντικά είναι η ταχύτητα με την οποία άλλες χώρες του κόσμου επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, ε, καταρτίζουν ε, μηχανικούς, κατακτούν τις αγορές και μερικές φορές παραβιάζοντας τους διεθνείς κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι το επικίνδυνο και αυτό θα είναι η κορυφαία μου προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κονέσκνα από την ΚΟΥ είναι η τελευταία ομιλήτρια του πρώτου γύρου των ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Οριστήσα Επίτροπε. Welcome. Uh, Θα ήθελα να πω ότι για μένα ε, είσαστε αξιοθαύμαστοι, διότι έχετε, ε, έχετε τον χρόνο να είσαστε και ευρωβουλευτή ε, και να έχετε δουλειά που να βγάζετε 10.000 ευρώ το μήνα. με όλη αυτή τη δουλειά που είχατε να κάνει για την ομάδα προβληματισμού αυτή, αυτού, αυτή, αυτό απαιτεί πάρα πολλά. εγώ δεν θα μπορούσα να ε, φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει δύο δουλειές πλήρους απασχόλησης ε, ταυτόχρονα με όλη τη δουλειά που έχω. Σας θαυμάζω λοιπόν γι' αυτό. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμήνης, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα σχετικά με τη διαδικασία, πώς θα διαμορφωθεί. τι μηχανισμούς ελέγχου μπορείτε να ε, διασφαλίσετε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμήνη. και η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με τον τουρισμό, διότι είσαστε αρμόδια και για τον τουρισμό, ε, που αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής διεύθυνση Ανάπτυξης, ε, DG Grow. Στην επιστολή της εκλεγής σας Προέδρου και ούτε στις απαντήσεις σας βρήκα ε, οτιδήποτε, κάποιο στοιχείο για τον τουρισμό. Ε, είχαμε άλλωστε και την υπόθεση Thomas Cook. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον ακούτε φοροτιμή στο πόσο δυναμική είμαι. Τώρα, για το θέμα τη αμυνά είναι πολύ σημαντικό όντω. Και πρέπει να σεβαστούμε όλε τι διαδικασίε και να ελεγχθούν η όλη διαδικασία ήταν συλλογική, ομαδική μάλλον, διότι βασίστηκε στην απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ομάδα εμπειρογνωμόνων που εξαρτώνται από τα κάτι μέλη. Στη φάση τη επιλογή ενό προγράμματο πρώτα και μετά ώστε να λάβουμε και τα εχέγγυα. Είναι ε, ομαδική δουλειά, ε, συλλογική διαδικασία, με διαδικασίε που είναι εντελώ αμερόληπτε. Ε, Εδώ η δική μου δουλειά θα είναι ανάλογη με αυτή και των υπόλοιπων επιτρόπων. Αυτό το ταμείο λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικό για να ενισχύσουμε μια σειρά από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επειδή η παγκόσμια ασφάλεια, ιδίω σε αυτή την χρονική στιγμή, απειλείται πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε διανοηθεί πριν από κάποια χρόνια. Γι' αυτό θα επενδύσουμε από κοινού σε αυτή την κοινή προσπάθεια η οποία υπάρχει. Ήδη έχουν επιχειρήσει επιχειρήσεις από τρία κράτη-μέλη. Εάν αυτό λοιπόν σας ανησυχεί ότι οι μεγάλε όπως λέγονται χώρες θα πάρουν όλες τη χρηματοδότηση, δεν είναι έτσι. Και θα συμμετάσχουν και άλλε μικρομεσαίες, πολλέ μικρομεσαίες. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι συμμετέχοντε, όμω η χρηματοδότηση θα πάει τι ευρωπαϊκέ εταιρείε και μπορούν οι φορολογούμενοι τη Ευρώπη να χαίρονται διότι θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Πώ μπορούν όλα αυτά να ελεγχθούν. Ήρθα εδώ για να σα μιλήσω. Εάν με εμπιστευτείτε και με εγκρίνετε, ε, λογικό θα είναι να έρχομαι συχνά για να συνομιλούμε κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα που αφορά ένα κάτω μέλο, και όταν ένα φάκελο, ένα θέμα περνάει από το κολέγιο των επιτρόπων θα μπορούμε να το συζητούμε. Είναι σοβαρό και είναι και απαραίτητο και δεσμεύομαι να το πράξω. Επερώτηση. Κυρία Κονέτσινα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, διότι δεν το αναφέρατε. Είναι κάτι που διαμορφώνει την εσωτερική αγορά, που κλονίζει την εσωτερική, την εσωτερική αγορά αυτή τη στιγμή, καθώς και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η ε, δημόσιες επιχειρήσεις ε, και οι διευθυντές τους ε, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι αρμοδιότητα πάντως της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Ναι, όντως ξέφυγα από το άλλο θέμα και άφησα τον τουρισμό. Ε, είμαι από την από, μάλλον γνωρίζω καλά μέρη όπω η Μασαλία στη Μεσόγειο και γνωρίζω πολύ καλά και τα θέματα του τουρισμού. Με φάνταστε ότι δεν με ενδιαφέρει. Είμαστε ο πρώτο παγκόσμιο τουρισμό, ε, ε προορισμό για τον τουρισμό, συγγνώμη. Η δημοκρατία τη Τσεχία το γνωρίζει αυτό πολύ καλά, δεδομένου του πόσο τη ομορφιά μια πόλη όπω η Πράγα. Ε, και βεβαίω δεν είναι μόνο αρμοδιότητα τη Γενική Διεύθυνση Grow, Ανάπτυξη αλλά και πολλών άλλων γενικών διευθύνσεων ταυτόχρονα. Πάντω εδώ μπορώ να σα δώσω την προσωπική μου άποψη. Η αηφορία είναι το βασικό εδώ. Πώ να βεβαιωθούμε ότι τόσο όμορφε πόλει, θαυμάσιε πόλει, νέε περιοχέ, ε, παραλίε δεν πέφτουν θύματα τη ίδια τη επιτυχία του. Είναι θέμα αηφορία λοιπόν εδώ. Και είναι και θέμα ανθρωπίνων πόρων. Διότι ο τουρισμό προκαλεί και έχει μεγάλη ανάγκη από εργατικά χέρια. Και υπάρχει και θέμα πλατφόρμα τι πλατφόρμες συνεργατικέ, σωματικέ, θα χρησιμοποιήσει κανεί για τι μεταφορέ για τι κρατήσει, διότι πρέπει να κοιτάξουμε οι δραστηριότητε των ανθρώπων, το πώ θα νοικιάζουν α πούμε τι κατοικίε του ώστε να δημιουργούν προβλήματα γειτονία τη πόλη να μην συνεχιστούν ανεξέλεγκτα. Ε, τα περιβαλλοντικά θέματα, η προστασία τη πολιτιστική κληρονομιά είναι πολλά θέματα λένετε εδώ και ελπίζω θα τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το πρώτο γύρο των ερωτήσεων και περνάμε στο δεύτερο γύρο τώρα ξεκινώντας από τον κύριο Τσεβε. Δίνω το λόγο στην κυρία Τεσούτερ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο λοιπόν, όπου τα μέλη διαφόρων επιτροπών θα θέσουν τις ερωτήσεις. Ένα λεπτό για την, απάν... για την πρώτη ερώτηση και ένα... λεπτό για την επερώτηση. Πρώτο ο κύριο Παύλο Αρία Ετσεβερία από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκουλάρ, όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτε ε, μα προειδοποιούν για μια νέα οικονομική ύφεση που κατά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων ίσως ε, έχει συνέπειες ε, σχεδόν ε, παρόμοιες με τις κρίσεις του 2009. Σήμερα ένας από τους μηχανισμούς που έχουμε για την απασχόληση δεν λειτουργήσε τότε ε, πλήρω λόγω του προστατευτισμού κάποιων κρατών μελών. Αυτόνομε μικρομεσαίε επιχειρήσει, επιχειρήσει ε, και καταναλωτέ υπέστησαν τα πάνδυνα λόγω αυτού του προστατευτισμού. Και ο προστατευτισμό αυτό ε, οδήγησε σε κάποιε θέσει ει βάρο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, νέου διοικητικού φραγμού και προβλήματα για βασικού. Τομεί τη ε, Ευρωπαϊκή Οικονομία, όπω είναι οι μεταφορέ και η μια αρχή τη ε, οικολογική ουδετερότητα. Και όμω αυτά είναι βάσει ε, τη εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά που συμπεριλαμβάνει και την ψηφιακή αγορά. Βέβαια, κατά μέσο όρο 8,4 μήνες χρειάζονται τα κρατημέλη για να μεταφέρουν τις οδηγίες του στο εσωτερικό δίκαιο. Θα προτείνεται σχέδιο δράση για να βελτιωθεί η εφαρμογή του ε, κοινοτικού δικαίου και να αποφύγουμε την στρέβλωση της ενίας αγοράς από εθνικά προστατευτικά μέτρα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκουλάρ, παρακαλώ. Κύριε ε, Βουλευτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί πραγματικά... Α, συγγνώμη, δεν μιλάω ισπανικά. Σας ευχαριστώ που μιλήσατε για το σύνδεσμο μεταξύ της μακροοικονομίας, δηλαδή την εξέλιξη των οικονομιών μας και τον πιθανό κίνδυνο ύφεση και του έργου της Επιτροπής σας. Ακριβώς τέτοια ε, νοοτροπία χρειαζόμαστε και τέτοια διαπαιδαγώγηση για τον κόσμο. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι για να αναπτυχθεί η ευημερία, κάτι που βέβαια είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής ΕΚΟΝ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να έχουμε εδώ ε, επιχειρήσεις που θα ευημερούν, ε, εύρυθμη λειτουργία, φιλοπεριβαλλοντική οικονομία και ούτω καθεξής. Για 18 μήνες εθήτευσε στην Τράπεζα της Γαλλίας και παρακολούθησε αυτό το θέμα το μακροοικονομικό εκ του σύνεγγης. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ε, ε, ανησυχίας, αλλά η ανωδική τάση του προστατευτισμού έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Και Όντω, κάποια μέτρα προστατευτικά μπορούν να μειώσουν την ανταγωνιστικότητά μα, αλλά μην ξεχνούμε ότι η οικονομία μα είναι τμήμα τη παγκόσμια οικονομία. Και ενδείξει ε, από χώρα όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν αλλάξει πορεία, ε, τον τρόπο που οι Κινέζοι αντιμετωπίζουν την ανάπτυξή του, το γεγονό ότι κάποιε χώρε λαμβάνουν ε, μέτρα αντιπερισπασμού ε, επίσης, ε, αν τελικά υλοποιηθεί το Brexit στα τέλη του μήνα, δεν ξέρω τι στρατηγική θα υιοθετήσει η Βρετανική κυβέρνηση. Οπότε έχετε δίκιο, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ενιαία αγορά. Και θα πρέπει από κοινού να εξηγήσουμε τα πλεονεκτήματα, κάνοντας και κάποιες θυσίες βραχυπρόθεσμα. Γιατί όταν κάνουμε μια, ένα συμβιβασμό, κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, αλλά έτσι θα εδραιώσουμε το περίπλοκο βιομηχανικό και κοινωνικό μας ιστό. Επίσης, έχουμε κάποιες εμπορικές συμφωνίες που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκι του Φιλ Χόγκαν, αλλά θα συνεργαστούμε στενά γιατί η αγορά έχει δύο σκέλη, εσωτερικό και εξωτερικό. Μέχρι στιγμής ε, ε, συγκεντρωθήκαμε υπερβολικά στις μεταξύ μας σχέσεις και δεν εξετάσαμε δεόντως πώς χρησιμοποιείται η αγορά και πώς απηχεί στις εξωτερικές μας σχέσεις επερώτηση από τον κύριο Τσεβαρία. Ευχαριστώ για την απάντηση. Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη προτιμούν τις περισσότερες φορές τις οδηγίες για λόγους που δεν έχουν σχέση με την εσωτερική ή την ενιαία αγορά. Εσείς δεσμεύεστε να χρησιμοποιείτε περισσότερο τους κανονισμούς που είναι καλύτερο μέσο εναρμόνισης της ενίας αγοράς από ότι οι οδηγίες. Στις γραπτές σας απαντήσεις είπατε ότι αν χρειαστεί θα λάβετε και πιο αυστηρά μέτρα, χωρίς να διστάσετε. Πώς θα προτείνετε πιο αποτελεσματικά μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των παραβιάσεων, ακόμη και μερικές φορές είναι πολιτικά αμφισβητήσιμες. Ευχαριστώ. Για το πρώτο θέμα, τι νομοθετικό μέσο θα επιλέξουμε, κανονισμό ή οδηγία. Η προσωπική μου προτίμηση είναι υπέρ λιγότερων κανόνων που θα εφαρμόζονται όμως παντού. Άρα είμαι περισσότερο υπέρ του κανονισμού, γιατί είναι άμεση εφαρμογή στα κράτη-μέλη, αποφεύγεται η προθεσμία μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και αποφεύγονται οι αποκλήσει στην εφαρμογή που λέμε, χαρακτηρίζουμε τον ωραίο λόγο, ε, όρο gold plating του κανονιστικού υπερθεματισμού. Το θέμα είναι ότι η οδηγία ε, επινοήθηκε για να αφήσουμε ελεύθερο πεδίο στην επικουρικότητα και να μπορούν οι, τοπικοί, οι περιφερειακοί ή εθνικοί νομοθέτες να προσαρμόσουν την οδηγία στις εσωτερικές τους συνθήκες. Και κάθε φορά χρησιμοποιούμε το καταλληλότερο μέσο, το καταλληλότερο νομοθετικό μέσο ανάλογα με το με το σκοπό μας. Και ακόμη και για τις οδηγίες, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να τις εφαρμόσουν και να τις μεταφέρουν στην εσωτερική του ενωμένη τάξη. Και αν ε, μου δώσετε την έγκρισή σας, θα, θα προσπαθήσω να συνεργαστώ και με τα εθνικά κοινοβούλια για να δούμε πώς θα εφαρμόζονται οι οδηγίες. Και ε, είμαι υπέρ ε, πιο στενού πιο στενή συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Γιατί το πιο σημαντικό, το καλύτερο μέσο είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Γκάιερ για ένα λεπτό. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα ε, του βοηθού σας. Παρουσιάσατε την υπόθεση αυτή ως καθαρό θέμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Ωστόσο, η έρευνα του Όλαφ συνεχίζεται και αν έχω ενημερωθεί σωστά, τότε την ημέρα που σας επέλεξε η κυρία Φόντερ Λάιεν ε, έκανε έρευνες εις βάρος σας η ε, γαλλική ε, αστυνομία. Γιατί και μάλιστα παραιτηθήκατε από Υπουργό Αμήνη για να μπορέσετε να ασχοληθείτε με την υπόθεση. Γιατί νομίζετε όμω ότι μπορείτε να είστε επίτροπο και όχι Υπουργό Αμήνη. Ευχαριστώ. Δεν ήμουν σαφή μάλλον στοιχεία και γεγονότα. Όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο το 2009, προσέλαβα τη βοηθό του προκατόχου μου. Κάτι κλασικό. Δεν είχα πολιτική εμπειρία, έρχομαι από την κοινωνία των πολιτών, ήμουν υπεύθυνη για ευρωπαϊκή οργάνωση ο άνθρωπο αυτό εργάστηκε για πέντε χρόνια σε όλη τη διάρκεια τη θητεία μου και Γενικό Γραμματέα του Ευρωκοινοβουλίο αποφάσισε να κάνει ε, έλεγχο ε, αναρρύθμι των εγγράφων τα οποία χορήγησα διότι μου ζητήθηκαν. Έτσι γίνονται στι διοικητικέ διαδικασίε και δεν υπήρχε καμία διάθεση εξαπάτηση εδώ, καμία πρόθεση τέτοια. Ε, στο τέλο τη πρώτη θητεία και αποφασίζοντα να μην κρατήσω αυτόν τον βοηθό επειδή η διοργάνωση του γραφείου μου δεν ήταν καλή, δεν είχα τελικά τοπικό βοηθό στο δεύτερο μέρο τη θητεία μου, στη δεύτερη θητεία μου. Και αποφασίσαμε να μην γίνει παρέτηση ή μάλλον να υπάρξει ένα φιλικό διακανονισμό, ο οποίο κράτησε λίγο παραπάνω από την προβλεπόταν, διότι το εργατικό δίκαιο τη Γαλλία προστατεύει του μισθωτού. Και δεν ήθελα να οργανώσω μια ολόκληρη διαδικασία απόλυσης. Οπότε ήταν δική μου πρωτοβουλία να μην παραμείνω στην γαλλική κυβέρνηση. Αυτό είχε να κάνει, όπως είπα και στον κύριο Μπελαμή, ε, με μία παράδοση, ένα έθιμο που τώρα δεν ισχύει πλέον. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Φαντάζεστε ότι και μπορείτε να το ελέγξετε αυτό που λέω, ότι θα με συνέφερε να μην είναι έτσι. Όμω δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Η έρευνα κράτησε δύο χρόνια και συνεχίζεται. Και αυτή τη όλα αυτό το ίδιο. Λοιπόν, είμαι σε ε, φάση να βρίσκομαι σε δίκη και σέβομαι τη δικαιοσύνη τη χώρα μου, σέβομαι τη δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σέβομαι και την απόφαση τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που αποφάσισε ότι μπορώ να παρουσιαστώ μπροστά σα. Κύριε Γκάιερ, ερώτηση. Μάλιστα. και εάν... Εάν ε, υπάρξει ε, τελικά ε, δίωξή σας, θα παραιτηθείτε από επίτροπος. Δεν μπορώ να απαντάω σε ερωτήσεις τελείως υποθετικές. Δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν πρόκειται να καταδικαστώ, είναι μία πιθανότητα αυτή. Αλλά σήμερα, μιας και τα γεγονότα έχουν περάσει από την κρίση του Ευρωκοινοβουλίου, το κοινοβούλιο στο οποίο εργάστηκα, που κοίταξε πώς εργάστηκε αυτός ο βοηθός. Θέλω να φύγω με το κεφάλι ψηλά. Και εάν μου δείξετε την εμπιστοσύνη σας, θα μπορούμε να συνεργαστούμε για πέντε χρόνια. Διότι αν γίνει το ανάποδο, όποιο ε, είναι σε κατάσταση να τον ε, περνάνε από κάποια ε, έλεγχο, κάποια δίκη θα καταργηθεί το τεκμήριο της αθότητας. Το τεκμήριο αθότητας είναι ότι όταν κανεί καταδικαστεί θα πρέπει να υποστεί τι συνέπειε. Όταν όμω καταδικαστεί, αν μου συμβεί, θα το κάνω. Αλλά τώρα είναι ακόμα υποθετικό το ερώτημα. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Φλέγκο. Εκ μέρου των του Renew, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Κουλάρ. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε υποψήφιο επίτροπος για το νέο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να βάλουμε νέα θέματα για την Ψηφιακή Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις πέντε προτεραιότητες ε, πέντε προτεραιότητες ψηφιακής Ευρώπης χρηματοδότησε 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού του ποσού, αν και το Συμβούλιο είναι υπέρ της περικοπής του προϋπολογισμού. Πώς μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε να ψηφιοποιήσουμε επιτυχώς την κοινωνία και τις επιχειρήσεις αν γίνουν περικοπές στον προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό της ψηφιακής Ευρώπης. Εσείς ως υποψήφια επίτροπος ε, θα ταχθείτε με πυγμή και απερίφραστα υπέρ της ισχυρής χρηματοδότησης του προγράμματος ψηφιακής Ευρώπης για το επόμενο ΠΔΕΛΤΑΠ 2021-2027 για να εξασφαλίσουμε επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ψηφιακή Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Φλέγκο. Κυρία Γκουλάρ. Περίμενα το τέλος της διερμηνίας για να μην χάσω κανένα κομμάτι της παρέμβασής σας. Πολύ σημαντικό το θέμα που θίξατε, γιατί αναφέρεστε σε βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναφυσβήτητα θα δώσουμε μάχη για να υπερασπίσουμε τον προπολογισμό, γιατί αυτό το κονδύλιο 9,2 δισεκατομμύρια για την επταετία 21-27, αν το συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα κονδύλια που οι ανταγωνιστές μας αφιερώνουν για τα ψηφιακά ζητήματα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι τόσο υψηλό. Φυσικά και θα δώσω μάχη για να παραμείνει ε, δαψιλής ο προϋπολογισμός του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Επίσης, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα εννοείται, ε, της τις δημοσιονομικές προοπτικές και το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα το διαπραγματευτούν τα κράτη-μέλη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σίγουρα το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν είναι και πολύ θετικό με περιθώριο λιγμό σχετικά περιορισμένο, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα προγράμματα να πείσουν για την ωφέλειά τους και τη χρησιμότητά τους. Και με τη συνεργασία μας, με τα ίδια ποσά, θα έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πιστούν ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουν από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα συνεργαστούμε και θα βάλουμε τα δυνατά μα για να υλοποιήσουμε το στόχο μα. Εγώ θα, πραγματικά θα δώσω μάχη ω να θα αγωνιστώ υπέρ τη διατήρηση του προπολογισμού, αλλά δεν ανήκει σε μένα τελική απόφαση για την κατανομή των κονδυλίων. Και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα στεγανά των διαφορών τομέων. Γιατί ο κάθε επίτροπο θα δώσει μάχη για το δικό του χαρτοφυλάκιο και σε τελική ανάλυση θα γίνει μία κατανομή και ένα συμβιβασμό. Εγώ φυσικά θα προτιμούσα να έχει υψηλότερε αρμοδιότητε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δημοσιονομικά ζητήματα. Γιατί έχουμε πραγματικά μία ξεχωριστή διαδικασία, μοναδική. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αντίστοιχε αρμοδιότητε στα θέματα αυτά με, το, με τα εθνικά κοινοβούλια που μπορούν να θεσπίζουν φορολογία και να έχουν έλεγχο το φορείς πρακτικών εσόδων. Κύριε Φλέγκο, έχετε επερώτηση. Όχι, δεν έχω επερώτηση. Θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω, κύριε Γκουλάρ, για την πολύ θετική ε, συγκεκριμένη και εύστοχη απάντηση. Σίγουρα η ψηφιοποίηση θα είναι στο μέλλον απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας και οικονομίας και για την ε, ποιοτική διαβίωση της κοινωνίας μας. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε υπέρ αυτού του σκοπού όλοι. Και κάθε γωνιά της Ευρώπης, από τη βορρά μέχρι ε, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, θα υποφεληθούμε από το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη στο μέλλον. Για όλου μα είναι σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Και για εσά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και για εμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για το Συμβούλιο, και για του επιχειρηματίε και για του καταναλωτέ. Γιατί οι καταναλωτέ και οι επιχειρηματίε περιμένουν από εμά απτά αποτελέσματα για τη βελτίωση τη καθημερινότητά του και του βιωτικού του επίπεδου. Σα ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Φλέγκο. Κυρία Γκουλάρ, έχετε κάτι να πείτε? Όχι. Δεν μπορώ να το πω στα Ογγρικά δυστυχώ, αλλά ευχαριστώ. Ο κύριος Ντιντιέ από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εκ μέρου του ΕΛΚ επιτρέψτε μου να ξαναπάμε στο θέμα του ρόλου σας στο Ινστιτούτο Μπέργκμαν. Δεν θέλω καθόλου να μαυρώσω την υπόλοιψή σας. Ούτε θέλουμε να αμφισβητήσουμε την ε, νομιμοποίηση κάποιου να έχει παράλληλες δραστηριότητες. Είναι θέμα ευθείας και δυναμισμού. Κοίτα, μας αρέσει είτε όχι, κανείς εδώ δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αιμοσύνη σας που δεν έχει τίποτα το τεχνητό. Εάν μου επιτρέπετε αυτήν την, ε, αυτόν τον αστεισμό, αφού θα αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου σας. Πάντως, αφού πρόκειται για ένα ποσό, ένα ποσό που είναι διπλάσιο αυτού του, το οποίο λαμβάνατε ως ε, ε, ευρωβουλευτής. Ήταν κατά την άποψή σας συνετό και η ερώτησή μου είναι σχεδόν προσωπική. Εάν ξέρατε ότι θα γινόσαστε κάποια μέρα Ευρωπαία Επίτροπος, θα το δεχόσαστε αυτό ε, το ποσό από αμερικανικές πηγές και ειλικρινώς εάν δείτε μέσα σας, αν έπρεπε να το ξανασκεφτείτε, θα το κάνατε όπως το κάνατε. Ε, ευχαριστώ κύριε Διδιέ. Ξέρω ότι είναι μεγάλα τα ποσά, είναι υπέροχα. Ε, και το έχω πει και στο κοινοβούλιο, δεν ξέρω πώ μεταφράστηκε και ακούστηκε, αλλά πολλά χρόνια ασχολήθηκα με την καταπολέμηση τη φτώχεια. Καταλαβαίνω. Έχω πολύ συχνά επαφή με ανθρώπου που δεν ξέρουν πώ θα κλείσουν το μήνα. Αλλά είναι λίγο τεχνητό να συγκρίνει κανεί ποσά. Νομίζω είστε δικηγόρο στο Δικηγορικό Σύλλογο τη Νέα Υόρκη. Σωστά. Ω τέτοιο, θα πρέπει να γνωρίζετε τι απολαυέ των Αμερικανών δικηγόρων θα ξέρετε τι χρεώνουν οι consultants, οι σύμβουλοι. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνουμε επαγγελματική δίκη εδώ, απλώς λέω να το έχουμε κατά νου. Και έχω συνέστηση ότι η ιδέα της συμμετοχής όλων, ότι όλο το κοινωνικό φάσμα πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχει, είναι μια προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια που επιτρέπει ε, ο κόσμος να αναπτύσσει διάλογο μεταξύ τους στο Ινστιτούτο Μπέργκμαν είχα διάλογο και συνομιλήσω με πολλούς Ευρωπαίους. Ήταν κυρίω Ευρωπαίοι τα μέλη εκεί που εγώ συμμετείχα, παρόλο που λέτε αμερικανικές πηγέ ή αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό που δεν ε, μετανιώνω είναι ο ενθουσιασμό που είχα όταν ανακάλυψα τη δράση αυτού του Ινστιτούτου να πω ότι «Α, για δε, κάνουν πράγματα συναρπαστικά». Συμβαίνει στη ζωή αυτό. Κάποιε φορέ στη ζωή μα, βρίσκουμε ότι κάποιο κάνει κάτι ενδιαφέρον και δεχόμαστε μια πρόταση όχι. Αυτό που μετανιώνω όμω είναι ο τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό σε σήμερα. Ε, είναι κρίμα που ε, βεβαίω κάνετε τη δουλειά σα, δεν ε, ασκώ κριτική εναντίον σα, αλλά είναι κρίμα που πέφτει αυτό το φως αυτή την υπόθεση. Και είναι κρίμα που πραγματικά κάποιοι εθίγησαν, κάποιοι ε, ίσως ε, τσουγκρίστηκαν στις ευαισθησίες τους με αυτή την υπόθεση. κάποιοι με ταλέντο ή νομοσύνη είναι κρίμα να μην μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Βέβαια, ίσως τα πράγματα να γίνονται και λίγο διαφορετικά. Και βεβαίω είναι προσωπικό το χρηματικό όφελο και βεβαίω τα συμφέροντα μπορεί να αμφισβητηθούν, όμω το ποσό είναι δηλωμένο. Αν είναι νόμιμο και δηλωμένο, γιατί να αμφισβητείτε ε, εφόσον δεν υπήρξε θέμα ελέγχου. Επερώτηση κύριε Τιντιέ. Ευχαριστώ. Διευκρινίζω εδώ ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ τη δική σα πορεία και τη δική μου. Εγώ στη σταδιοδρομία που αποφάσισα τη μέρα που έγινε Ευρωβουλευτή να διακόψω οποιαδήποτε δραστηριότητα που είχε σχέση με αμερικανικά συμφέροντα και διέκοψα την δραστηριότητά μου ω δικηγόρο στον Δικηγορικό Σύλλογο τη Νέα Υόρκη. Ο καθένα μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όμω αυτό ε, είναι άλλο θέμα. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι στα πλαίσια τη δραστηριότητα που είχατε αναπτύξει στο Ινστιτούτο των Μπέρμαν δεν χρησιμοποίησατε ποτέ πληροφορίε εμπιστευτικέ τι οποίε θα μπορούσατε να έχετε γνωρίσει, να έχετε μάθει ω ε, ε, ευρωβουλευτή ή έχοντας επαφή με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κυρία Γκουλάρη. Σας το διαβεβαιώ. Δεν είναι εκτελεστική η δουλειά του Ευρωβουλευτή ούτε έχει πρόσβαση σε απόρριτε πληροφορίε. Είναι διαφανέ στο σώμα μα. Όλε οι αποφάσει που παίρνουμε είναι διαφανεί. Και εργαζόμαστε σε ομάδε ευρωβουλευτών. Είχα την τύχη να εργαστώ με πολλού από εσά, με την Ελίζα Φεραίρα, ε, χάρη, που επίση θα γίνει, τέλο πάντων, ε, αν όλα πάνε καλά, εξίσου καλά θα τα πάει και εκείνη, εφόσον εγκριθούμε και οι δύο. Αλλά πάντοτε συνομιλούσαμε μεταξύ μα. Κανεί δεν είχε πρόσβαση σε κάτι που θα μπορούσε αυτό καθε αυτό. Όταν κανεί υποβάλλει τροπολογίε, είναι ένα άνθρωπο, ένα άτομο, μια φωνή, μια ψήφο. Ε, όλη η διαδικασία ε, οικοδόμηση, χτισήματο τη νομοθεσία είναι ομαδική. Δεν είχα πρόσβαση σε μυστικέ απόρριτε πληροφορίε. Δεν ε, είχα περισσότερη πρόσβαση από έναν κλασικό εισηγητή. Με αυτά και με αυτά λοιπόν μπορώ να πω ότι δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί τέτοιο πρόβλημα και το λέω ειλικρινώ. Δεν θα το έκανα εφόσον είχα κάποιο εκτελεστικό λειτουργήμα νομοθετικού χαρακτήρα. Ευχαριστούμε κυρία Κέπχαρτ εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Σας ευχαριστώ κυρία Κουλάρ. Ειλικρινά πρέπει να πω ότι ακόμη δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσατε να παραμείνετε ε, υπουργό στη χώρα σας ε, λόγω της έρευνας ε, εις βάρος σας. Ε, πιστεύετε όμως ότι μπορείτε να είσαστε επίτροπος είπατε ότι θα ανοίξετε πάλι τη συζήτηση για τις υπηρεσίες. Μετά από μακρά συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και με το Συμβούλιο, ε, βρήκαμε μια συνενετική λύση ε, για την πρόταση αυτή για τις υπηρεσίες. Αλλά εσείς θέλετε πάλι να ξανανοίξουμε το θέμα, να έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα στα συστήματα ασφάλισης στα διάφορα κρατημέλη. Πώς να ερμηνεύσω αυτό που είπατε. Η κυρία Γκουλάρ, παρακαλώ. Καταρχήν, κυρία Γκέπχαρτ. Δεν ήμουνα στην ίδια θέση τον Ιούνιο του 2017. Ούτε τις ίδιες αρμοδιότητες είχα. Δεν υπήρχε το θέμα της εμπλοκής των στρατευμάτων τότε και το μόνο που μπορώ να σας πω και τότε σας κατάματα είναι ότι τότε, το 2017, δεν ένιωσα α, σε θέση να πω θα αφήσω τα στρατεύματα που βρίσκονται επί τόπου στην επιχείρηση Φρουρός. Είναι θέμα προσωπικό, εσείς μπορεί να διαφωνείτε. Σας είπα τότε πώς ένιωσα, το 2017. Δεύτερο, δεύτερη ειδοποιώς διαφορά με την σημερινή διαδικασία είναι ότι έδωσε εξηγήσει, η διαδικασία έχει προχωρήσει και δεν πρέπει φυσικά να προδικάζουμε τίποτα γιατί το θέμα βρίσκεται στο δικαστήριο και μετά την ε, κατάθεση που έδωσα δεν τέθηκα υπό έρευνα. Και εσείς θα κρίνετε αν ε, αυτά αρκούν ως εξηγήσεις. Δεν είναι δική μου επιλογή η αρμοδιότητα, αλλά είναι σημαντικό να τα υπενθυμίσουμε όλα αυτά. Επίσης, ποιος είναι ο στόχος για τις υπηρεσίες. Στόχος δεν είναι η απελευθέρωση Γι' αυτό είπα προηγουμένως, η... δεν είναι αυτός σκοπός η απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών. Στόχος είναι να μπορούμε ταυτόχρονα, και γι' αυτό το επισήμανα προηγουμένως, η, οικονομία, η κοινωνική οικονομία, δηλαδή ο συνδυασμός ε, του οικονομικού με το κοινωνικό σκέλος. Και να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές ε, ανταλλαγές και οικονομία, και ταυτόχρονα να σεβαστούμε τα κοινωνικά ζητήματα. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έχουμε ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Και όπως είπε ο κύριος Ετσαβαρία, έχουμε μια κατάσταση α, κινδύνου. Βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη συγκυρία, οπότε θα πρέπει να αναζητήσουμε θέσεις απασχόλησης, αλλά όχι πάση θυσία, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Και περίεργο, εγώ περίμενα ερωτήσει από εσά για τη θέσπιση του κατώτατου μισθού. Περίμενα από εσά ερωτήσει για την καταπολέμηση τη φτώχεια. Και αυτά βρίσκονται στο πρόγραμμα τη κυρία Φοντερ Λάιν, κυρία Γκέπχαρτ. Κυρία Γκέπχαρτ, για περώτηση. Ε, τέτοια θέματα αφορούν μια άλλη αντιπροσωπεία, την ε, Επιτροπή Απασχόλησης, ε, αλλά, εν πάση πτώση, Ακόμη δεν καταλαβαίνω την διατύπωσή σας για νέο άνοιγμα των συζητήσεων για τις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, θα προτείνετε οδηγία ή κανονισμό όπου θα λαμβάνετε υπόψη το εργασιακό δίκαιο Ε, στην ε, οικονομία αυτή της πλατφόρμας όπως ονομάζεται. Ναι ή όχι. Ωραία. Okay. Kurz Πολύ σύντομα, ναι. Θα πρέπει να δώσουμε σημασία στις νέες αυτές πτυχές της οικονομίας μας θα πρέπει να φροντίσουμε όχι να τις ελέγξουμε, αλλά να εξετάσουμε προσεκτικά τι ακριβώς γίνεται εκεί και οι εργαζόμενοι στους τομείς αυτούς ε, να προστατεύονται. Είναι σημαντική η προστασία. Δεν μπορώ να σας δώσω σήμερα πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες. Ε, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ βιαστικό. Θα πρέπει να συνομιλήσω με τους συνεργάτες μου. Ε, εάν ε, όμως ε, επιβεβαιώσετε τον διορισμό μου, εγκρίνετε τον διορισμό μου, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Από τους πράσινους ο κύριος Μπλος. Και άλλο ένα σημαντικό θέμα για πολλούς πολίτες. Για το Dieselgate, το σχετικό σκάνδαλο. Εκατομμύρια οχήματα στους δρόμους της Ευρώπης και 500.000 ε, απώλεια ετησίω με τεράστιες, ε, τεράστιους όγκους του άνθρακα εκπομπές. Μεγάλη ζημιά για την Ευρώπη. Και αυτό γιατί δεν ανακλήθηκαν εγκαίρω τα οχήματα, αλλά οι καταναλωτέ βρέθηκαν εξαπατημένοι να ψάχνουν αποζημιώσει. Θα πρέπει τέτοιε διαδικασίε να προβλεφθούν, ώστε το, η, Επιτροπή να αξιοποιήσει και τι ε, υπηρεσίες για να υποχρεωθείτε, σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις, να αναλάβετε και μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, κάποια κράτη-μέλη έχουν δώσει διαφορετικά όρια για τις άδειες εκπομπών αριών του θερμοκηπίου στο 2050. Πώς θα υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη που έχουν σκοπό να περιορίσουν αυτές τις εκπομπές σημαντικά. Κύριε Γκουλάρ, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρόκειται για ένα θέμα σημαντικό εξαιτία της ρήπανση και των συνεπειών που έχει στην υγεία. Και στην υπόθεση αυτή υπήρχε ένα στοιχείο εξαπάτηση των καταναλωτών. όντω ε, τους ξεγέλασαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοίταξε πώς μπορεί να βελτιώσει τους κανόνες, όχι να κάνει τι ίδιε τι δοκιμέ, να βελτιώσει τι συνθήκε ε, εντός των οποίων διοργανώνονται οι δοκιμέ με ένα σύστημα θα έπρεπε να έχει και νέες αρμοδιότητες. Αλλά εξαντλήσαμε νομίζω τις αρμοδιότητες που υπήρχαν. Δεν ξέρω να σας πω σήμερα πώς ακριβώς. Διότι θα πρέπει να το δούμε και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που τώρα για κάποιε συγκεκριμένε περιπτώσει είναι κάπω επιφυλακτικά. Δεν κάνουν και ό,τι περνάει από το χέρι του. Πρέπει όμω να βεβαιωθούμε ότι στην πράξη, στην πραγματικότητα, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δεν ήρθα εδώ να σα πω ότι υπάρχει η τέλεια λύση, η απόλυτη συνταγή και ότι μόλι έρθω στι Βρυξέλλε ε, θα μεταπίσω τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν είναι θέμα πίεσης της κοινή γνώμης, είναι θέμα πίεσης ε, μόνο των ιδίων ως ερετών αντιπροσώπων ε, στους εθνικούς ασφορεί. Ξέρω ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν κόμματα που ασκούν πίεση. Πρέπει οι εταιρείε, οι βιομηχανίε, να μην είναι πλέον σε θέση να εξαπατήσουν ή να διοργανώσουν ένα τέτοιου είδους κόλπο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει λίγο να πάμε παραπίσω και να πούμε ότι το δικαίωμα επιβολής ποινών πρέπει να ε, χρησιμοποιείται και να ασκείται οποτεδήποτε χρειάζεται χωρίς να υπάρχει δισταγμός. Όταν κάποιος αλλάξει την στάση του πρέπει να το κάνει εγκαίρος. Ιδάλλως βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μπορεί να παίξουν ασφαλιστικά μέτρα και αυτό να πάρει καιρό. Αν όμως χρειαστεί θα εξαντλήσουμε το πλωστάσιο που διαθέτουμε. Κύριε Μπλός, επερώτηση. Ναι, μιλήσατε για νέους κανόνες και επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία. Όμως υπάρχουν οριακές τιμές που ξέρουμε ότι έχουν, ε, τις έχουν υπερβεί οι εταιρείε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει δικασία επιπαραβάση και ένα σύνολο ερωτήσεων. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσάς. Εσείς δεσμεύεστε αυτήν τη νέα, ε, ε, αυτό το νέο θέμα να εξετάσετε αυτό το νέο θέμα και την, ε, ε, να διαμορφώσετε αναλόγως την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τι θα κάνουμε ε, αν η Γαλλία ας πούμε, από το 2050 μπορεί να διοδοτεί μόνο νοχήματα απαλλαγμένα τελείως από εκπομπές. Η Γαλλία έχει κάνει μια πολύ θετική ανακοίνωση, αλλά εσείς πρόκειται να υποστηρίξετε άλλα κάτι μέλη για να λάβουν τέτοια μέτρα συνολικά στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρ. Για το θέμα εφαρμογής του δικαίου. Δεν ε, πρόκειται να. Θα το επαναλάβω μάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξαντλήσει ό,τι εργαλείο έχει στα χέρια της. Δεν υπάρχει εδώ αμφιβολία. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Εάν τώρα θεωρείται σε κάποιες χώρες υπάρχουν νομοθεσίε που είναι πιο προηγμένε, πιο προχωρημένες, Πρέπει να το σκεφτεί κανεί προ στιγμή. Δεν έχω κάποια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται με την κάθε νομοθεσία ξεχωριστά. Δεν είμαι ειδική. Ξέρω τη γαλλική νομοθεσία, αλλά όχι ω εμπειρογνώμων. Τώρα, αν χρειαστεί να αποσύρουμε κάποιο κείμενο, λέτε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποσύρει πρόταση, αν χρειαστεί. Αλλά πρέπει να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά. Διότι κάθε κείμενο είναι καρπό δουλειά. Το ερώτημα είναι αν μπορεί κανεί να κάνει κάτι καλύτερο. Εάν ένα κείμενο μπορεί να φτάσει σε κάποιο αίσιο πέρα, είναι κάτι. Αν μπορεί να τροποποιηθεί και να γίνει καλύτερο, και αυτό είναι σημαντικό. Σε κάποια νομοθετική διαδικασία θυμάμαι ότι είχαμε ζήσει το να μεταβάλλονται δραματικά τα κείμενα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν υπήρχε ανάγκη απόσυρση. Είχαν ήδη μεταμορφωθεί. Οπότε θα είμαι ρεαλίστρια, θα εξαντλήσουμε όλα τα εργαλεία και θα δούμε όταν θα έχουμε πάει λίγο παραπέρα στην εξέταση του θέματο. Ο κύριο Θιερή Μαριανή από την Ήτρε. Ευχαριστώ. Κύριε Αγκουλάρ, Η Επιτροπή Γιούρι, όπω είπατε, νομικών υποθέσεων που διερευνά σύγκρουση φερόντων, όντω επικύρωσε την υποψηφιότητά σα αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω υπό ποιους όρους το έκανε. Ενώ υποψήφιος επίτροπος ε, ε, ε, έχουν απορριφθεί δύο Ρουμάνε και ο Ούγκρος, γιατί υπήρχαν υπόνοιες για τη σύγκρουση φερόντων. Στη δική σας περίπτωση επετράπει η διοργάνωση ακρόασης παρά το αντίθετο αίτημα του Ζήλου Μπρετών. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπατε, ήσασταν ε, λαμβάνεται αμοιβή από το Ινστιτούτο Περγκρουέν που υποτίθεται έχει φιλαθροφικό χαρακτήρα αλλά όχι και ανιδιοτελή. Ο, χρη, ο δισεκατομμυρίουχος που χρηματοδότησε αυτό το Think Tank έχει πολλές α, ε, οικονομικές δραστηριότητες. Μια και το ξέρετε και σας υποστηρίζει, μάλιστα μας έστειλε και επιστολή σήμερα το πρωί, ποιες είναι οι δραστηριότητες ε, του δισεκατομμυρίουχου που χρηματοδοτούν αυτό το Ινστιτούτο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο οποίο απασχοληθήκατε κι εσείς και λαμβάνατε και αμοιβή. Με Σε ό,τι αφορά την απόφαση Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Γιούρη δεν θα εκφέρω εγώ κρίση. Δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι διαδικασία, μάλιστα πρόσφατη διαδικασία που θεσπίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν ε, κρίνεται κάτι αδικαιολόγητο ή κάποιε παρατυπίε ή ατασταλίε, ε, δεν είναι δεν είναι δικό μου έργο να το σχολιάσω. Σε ό,τι ε, σε ό,τι αφορά την αμοιβή, είπατε ότι με απασχόλησε, ήμουν μισθωτή στο Ινστιτούτο Μπεργκουρέν. Όχι, ήμουν σύμβουλος, δεν είναι το ίδιο ε, νομικά. Επίσης, ε, δεν έχω ιδέα για τις ε, δραστηριότητες, οικονομικές δραστηριότητες του Διευθυντού του Ινστιτούτου. Εγώ ε, γνωρίζω μόνο τις δραστηριότητες του Think Tank. Ο Νικολά Μπεριό βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον, ε, μια ενδιαφέρουσα πορεία. Βέβαια και εσείς ε, διατελέσατε υπουργό, γνωρίζετε καλά τα πράγματα και σέβομαι τον τρόπο που αντιμετωπίζετε και τη θεώρησή σας. Είπατε ότι από τη στιγμή που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα αυτό το Ινστιτούτο σίγουρα κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Εγώ διαφορετική αίσθηση έχω. Ο Νίκολα Μπέργκριν ήταν, ε, είναι γιος του Χάινς Μπέργκριν ε, που ήταν Γερμανός που διώχθηκε από τους ε, Ναζί. Εξορίστηκε, έφυγε από την Γερμανία και ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα Μαντλέν Ολμπράιτ έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και είναι πολλοί οι Αμερικανοί που πραγματικά προβληματίζονται και ανησυχούν για αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Και γι' αυτό με τον Αμερικανικό τρόπο αναπτύσσουν κάποιε ιδέε ανάλογα με τι πεπιθήσει του. Μπορεί να μην τι ημερίζεστε, να μην τι εστερνίζεστε. Είναι δικό σα θέμα. Πάντω, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κάποιες ιστερόβουλες σκέψεις, αλλά ανάλογα με την πορεία τους ακολουθούν τις πεπιθήσεις τους. Είναι ο Νικολά Μπερκριν ε, ένιωσε την ανάγκη με βάση το παρελθόν του και την προέλευσή του έκρινε σκόπιμο να στήσει αυτό το think tank και να συμβάλλει στη βελτίωση του κόσμου. Και ναι, δεν νομίζω ότι ήταν επιλήψιμη αυτή η συμμετοχή μου. Μα δεν ε, λιδωρώ κανέναν, κυρία Γκουλάρ. Απλώς ο κύριος Νικολά Μπεργκρουέν είναι ο πρώτος χορηγός του Ινστιτούτου Μπεργκρουέν στο κέντρο της Κίνας για την τεχνητή νομοσύνη και ως insider των επιχειρήσεων έχει επενδύσει τεράστια ποσά στην Καλιφόρνια στηρίζοντας επιχειρήσεις. Επίσης, 25 εκατομμύρια έδωσε στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Είναι γνωστός ανταγωνιστής λοιπόν ε, της ενιαίας αγοράς. Μάλιστα, ε, φέτος ε, εξαγόρασε την ε, μεγαλύτερη εταιρεία ειδικών μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι έχει συμφέροντα ο Νικολά Μπεργκρόν. Και είπατε ήσασταν σύμβουλο. Σίγουρα έχετε προνομιούχες σχέσεις μαζί του. Αυτό δεν επηρεάζει τον τομέα που είναι το χαρτοφυλάκιό σας, γιατί είστε ε, η θεματοφύλακας ε, του ευρωπαϊκού τομέα. Και όμως ε, οι επιχειρήσεις που θα ελέγχεται θα έχουν ανταγωνιστική σχέση με τον, τις επιχειρήσεις αυτού του ανθρώπου. Όσοι με γνωρίζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι δεν είμαι ευεπηρέαστη. Βέβαια, ο καθένα έχει τη γνώμη του για μένα, είναι προσωπικό το θέμα. Και κύριε Μαριανή, εσείς, μπορεί, εσείς μπορείτε να πιστεύετε ότι ο καλύτερος τρόπος να προστατευτείτε από, τη Κινέζικη, από τον Κινέζικο ή τον Αμερικανικό ανταγωνισμό είναι να μην έχετε καμία σχέση με ε, τις χώρες αυτές ή εκπροσώπους τους. Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Και κυρίως για τα ψηφιακά ζητήματα, κυρίως για τα θέματα οικονομικής ανάπτυξης, η ζώνη Ασίας και Ειρηνικού είναι πολύ σημαντική. Και αν μου την έγκρισή σας, Φυσικά θα τηρήσω πιστά τις συνθήκες που απαιτούν ανεξαρτησία των επιτρόπων απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα και τα κράτη-μέλη, αλλά φυσικά έχουμε όλοι επαφές και δεν υπάρχει λόγος για να τις κατηγορούμε ή να δαιμονοποιούμε ορισμένες από αυτές. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κρασνοντέμσκι από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κύριε, κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και άλλες επιχειρήσεις ε, σε σχέση με τον τομέα αμήνης. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, τι συγκεκριμένα βήματα θα αναλάβετε ώστε να επιτρέψετε διευρυμένη συνεργασία διασυνοριακή ανάμεσα σε νομικά πρόσωπα. Ε, υπάρχουν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις αμήνης που ε, συνεργάζονται διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια. Τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς για να αλλάξει ο αμυντικός τομέας le a Το Ταμείο έχει όντως ως στόχο να επιφέρει κάποιες αλλαγές. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά και ε, η κυρία Μπιενκόφσκα το σχεδίασε και μαζί της το συμφωνήσατε. Δεν ε, το θέσπισε εγώ. Παρ' όλα αυτά το στηρίζω και στόχο του, στόχος του Ταμείου είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και όρος που θέτει για τη χορήγηση των κονδυλίων, των πιστώσεων, είναι ε, όροι που ως προαπαιτούμενο θέτουν τη συνεργασία. Γιατί απαιτεί να ε, συμμετέχουν τουλάχιστον τρει επιχειρήσει από τρει διαφορετικέ χώρε για να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση ένα σχέδιο. Αυτό θα δημιουργήσει ένα δυναμισμό και ε, ενάβσματα σε συνεργασία. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται να γίνει εν μία νυχτή. Θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες, να συμμετέχουν ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενδεχομένως, νεοφύης επιχειρήσεις και δεν ξέρουμε υπό ποιους όρους ε, θα εγκρίνονται τα σχέδια, αλλά ο όρος είναι να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις χώρες τουλάχιστον τρει επιχειρήσεις από διαφορετικέ χώρε και η απόφαση θα λαμβάνεται συλλογικά. Οπότε δεν θα κάνουμε δίκη προθέσεων για το ποιον θα ευνοήσουμε τον ένα ει βάρο του άλλου. Κάποιε χώρε έχουν πιο ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία από άλλε. Αναφερθήκατε όμω στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ακριβώ επειδή μιλούμε για νέα θέματα, μπορούμε να κάνουμε μια ανακατανομή και να δώσουμε περισσότερη πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Τσεχία και η Σουηδία, παρόλο που δεν έχουν ανεπτυγμένο αμυντικό κλάδο, είναι απόλυτα ε, επιλέξιμες να συμμετέχουν. Γιατί όχι δεν πρόκειται να ευνοηθεί η Γαλλία. Τώρα, για τα διάφορα υλικά, για τα μη επαδρομένα αεροσκάφη κτλ. Όλα αυτά είναι ανοιχτά και η πρόσβαση ανοιχτή προς όλους. Ο κύριος Κρασοντέμσκι για επερώτηση. Θα συμφωνήσετε τότε με την γνώμη της Επιτρόπου Διανκόφσκα που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ την προηγούμενη εβδομάδα ότι Εάν τελικά οι δύο-τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, στον αμυντικό τομέα της Ευρώπης επωφεληθούν, δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μετά το 2027. Ναι, αλλά εάν στην, ε, στο κείμενο της Επιτροπής λέει τρία, εννοεί τρία. Okay. Thank you. So, thank you very much. Um, we'll go to the next. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Ζαμπίνε Φερχέιν από την Επιτροπή Κάλτ για το ΕΛΚ. Κυρία Γκουλάρ, ε, έχετε πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο. Σήμερα μάθαμε ότι ήδη στο παρελθόν κάνατε πολλά πράγματα ταυτόχρονα μπορείτε να διασφαλίσετε η πολιτική για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λάβει την προσοχή που απαιτεί, διότι είναι ένα από τα πιο πολύπτυχα θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθείτε και αν ναι, ποιες θα είναι συγκεκριμένα οι προτεραιότητές σας στον τομέα αυτών δεδομένης της διτή φύσης ε, του τομέα αυτού που ξεπερνάει ε, τους προβληματισμούς που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά. Πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με, τους, με τις άλλες ε, αρμόδιες επιτρόπους, την κυρία Γιούροβα και την κυρία Καπριέλ πώς μπορείτε να διασφαλίσετε μία ενιαία προσέγγιση στην διαμόρφωση πολιτικής για τα μίδια και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε την συνέπεια στο πρόγραμμα ανάμεσα στο πολιτιστικό και ε, το τμήμα του προγράμματος και το τμήμα που σχετίζεται με τα μίδια. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε τη συνοχή στο πρόγραμμα αυτό. Ναι. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά πολλές φορές οι γυναίκες είναι καλύτερα σε θέση να το πετύχουν αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω είναι να θέσω προτεραιότητε, αλλά όχι να δώσω την εντύπωση ότι προτιμάω ένα θέμα σε σχέση με κάποιο άλλο. Είναι πολύ ευρύ και επικύλωτο το χαρτοφυλάκιο. Σαφώς. Το καταλαβαίνετε. Έτσι το αντελήφθη η κυρία Φοντερ και θέλησε να μου το αναθέσει. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε με ευθεία να τα διερευνήσουμε σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Όλα αυτά που είναι βιομηχανία και πολιτισμός. Μια, μια κοινωνία στέκεται στα πόδια τη όταν έχει οικονομία που παράγει αγαθά, αλλά έχει και δυνατότητα σε πολιτιστικό επίπεδο να παραμένει ανοιχτό ανοιχτόμυαλη, να εμπλουτίζεται για να ανανεώνεται και να είναι ζωντανή. Είναι πολύ δυναμική η κοινωνία μας στην Ευρώπη, στην, στα θεάματα, στον κινηματογράφο, σε πολλά πράγματα. Μια οικονομία όμως που περνάει από το στάδιο της ψηφιοποίησης, με νέες πλατφόρμες, μπορεί να παραμείνει σε θέση πρωταγωνιστή, και στις υποθέσεις τις πιο προηγμένες όπως η τεχνολογία αλλά και σε θέματα όπως ο πολιτισμός. Εγώ λοιπόν πάντοτε θα έχω στραμμένο το βλέμμα διότι ο πολιτισμός πιστεύω παθιάζει και το ανθρώπινο «ον» θα, και θα έχω το βλέμμα στραμμένο και προς την κυρία Γκάμπιλ και τις, δικής, της αρμοδιότητες γιατί νομίζω ότι έχουμε κοινού χώρους δράσης θα κοιτάξουμε δημιουργική, με δημιουργική, πρωτοβουλίες για δημιουργική Ευρώπη, για την δημιουργικότητα να προάγουμε ε, και τη διάσταση αυτή που πιστεύω ότι θα ενδιαφέρει και το Ευρωκοινοβούλιο. Και σε συνεργασία με την κυρία Γιούροβα, το είπα και νωρίτερα ε, και σε σχέση με τους εκφράσεις μίσους είναι η πολυφωνία, η ποικιλομορφία στα μέσα μαζικής ενημέρωση, η ελευθερία έκφραση. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα ακριβώς πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες μεταξύ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως ελπίζω ότι θα εργαστούμε ως ομάδα στο δυνατόν αποτελεσματικότερα. Ευχαριστούμε κυρία ε, Φερχάιν. Επερώτηση. Ρωτώ συγκεκριμένα όσον αφορά την πολιτική για τα οπτικοακουστικά μέσα. Όπως γνωρίζετε, η ε, αναθεωρημένη οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες ε, που τέθηκε σε ισχύ από τα κράτη-μέλη ήταν ε, μια από τις πιο σημαντικές νομοθετικές πράξεις της θητείας μας. Το καθεστώς που δημιούργησε η οδηγία αυτή και που κρίθηκε επαρκές σε τις δύο τελευταίες ε, δεκαετίες αποτέλεσε τη βάση για την αναθεωρημένη οδηγία. Εσύ, εσείς σε τι θέση έχετε στο θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ξεκινήσει τώρα η επικείμενη αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ναι, δεν πρόκειται να αμφισβητήσω την αρχή που, έχω, έχουν θεσπίσει οι συνομοθέτες για την ευθύνη, το liability. Τώρα, αν κάποιε πτυχές ε, μπορούν να συζητηθούν και είμαι ανοιχτή στη συζήτηση, αφού ε, κάνουμε διαβουλεύσει με τους ενδιαφερομένους και συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με τις ακροάσεις αυτές ε, δεν προλάβαμε να συναντηθούμε καθόλου. Μια φορά βρεθήκαμε μόνο στο Ζαμβάλ, η υποψήφια επιτροπή. Εκεί γνωριστήκαμε και μιλήσαμε για γενικά θέματα. Δεν μπορώ λοιπόν να το διαθετήσω μόνη μου, γιατί είναι ζήτημα που άπτε πολλών αρμοδιοτήτων και χαρτοφυλακίων. Σε ό,τι αφορά την οδηγία που μεταφέρθηκε πέρυσι στα εσωτερικά δίκαια, θα πρέπει να αφήσουμε κάποιο χρόνο για να δούμε τα αποτελέσματα εφαρμογής της. Ακόμη δεν στέγνωσε το μελάνι της οδηγίας, δεν έχει μεταφερθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε την ευκαιρία να ελέγξουμε πώς θα γίνει η εφαρμογή. Πρώτα να δούμε πώς εφαρμόζεται μια δίκη και μετά χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις ή τροπολογίες. Ο κ. Κάρλος Κίντ, ο επόμενος ομιλητής από το Renew Europe. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκουλάρ, ξαναείπατε ότι είστε ταγμένοι στον ευρωπαϊκό σκοπό ε, και το δείχνουν και τα γεγονότα. 8 χρόνια Ευρωβουλευτής, 4 χρόνια ε, και είσαστε και ομα... Ε, πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ο ρόλος των επιχειρήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τη συμμετοχή όλων και την δημιουργία πλούτων, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και τις πραγματικέ τους ευθύνες. Τον περασμένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε ειδικά μέτρα για όσα προβλέπονται τώρα ε, για τις επιχειρήσεις με βασικό στόχο την κοινωνική ε, ένταξη και την συμμετοχή των ανθρώπων με αναπηρίες. Μπορείτε να μας πείτε τι έχετε κάνει και τι θα κάνετε μάλλον για να υποστηρίξετε τις επιχειρήσεις αυτές της κοινωνικής οικονομίας και να δώσετε δυνατότητες που προβλέπονται και στην Οδηγία 2014 για τις δημόσιες προμήθειες να προσαρμοστούν κάποιες τις δημόσιες προμήθειες αυτές τις ε, κοινωνικές επιχειρήσεις με τέτοια διάσταση. Ευχαριστώ κύριε Καρλ Είναι ένας ε, κόρος, ένας κλάδος πολύ σημαντικός και το αντελήφθην όταν εξελέγει. Διότι πραγματικά ε, οι κοινωνικές επιχειρήσεις με διάσταση αλληλεγγύης προσφέρουν απασχόληση σε ανθρώπους που για λόγους, λόγω των δυσκολιών της ζωής ή λόγω της απόστασης από μεγάλα αστικά κέντρα δεν είναι σε θέση να δουλέψουν στις ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις όπου τα πράγματα είναι και καλύτερα αμοιβόμενα. Σε κοινωνική λοιπόν ε, προοπτική τα πράγματα πάνε καλά και επιτρέπουν οι επιχειρήσεις αυτές να μένει ζωντανός ένας ιστός στο επίπεδο των απλών ανθρώπων. Ξέρω ότι η κυρία Τόγια στην Ιταλία δραστηριοποιείται σχετικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μένουμε κοντά ε, στο τι συμβαίνει στην πράξη, στο επίπεδο το ατομικό. Και ο πράσινος ε, το τομέα του πρασινίσματο είναι πολύ σημαντικό για αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυκλοφορία και οι μεταφορέ, η μείωση κατανάλωση κάποιων προϊόντων, η κοινή χρήση, η κοινοκτημοσύνη κάποιων αγαθών. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά. Και βλέπει κανεί έτσι ότι παλιώνει. Όταν ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο, ιδίω στην πρώτη μου θητεία, θυμάμαι ότι κάποια θέματα συζητιόνταν πολύ. Έκτοτε άλλαξαν οι προτεραιότητε. Ε, Άλλε πήραν την πρωτοκαθεδρία. Εδώ λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε για τις δημόσιες προμήθειες που αναφέρατε, πολύ σημαντικό. Οι δημόσιες προμήθειες, όπως υπόθηκε, πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλά στι δημόσιε προμήθειε είναι δύο τα μέρη, δύο πλευρέ. Είναι αυτό που αναθέτει τη σύμβαση και είναι και αυτό που ε, ε, κάνει την υποβάλλει υποψηφιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποχρεώσει αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, ε, αρχέ φορεί να διαλέξουν μια επιχείρηση βάρο κάποια άλλη. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα είναι χρησιμότερο φυσικά οι προμήθειε να είναι πρασινότερε, αλλά θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Ευχαριστούμε για την επερώτηση, ο κ. Καλεσκίνη. Ναι, για το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι το καταστατικό των επιχειρήσεων αυτών είναι πολύ διαφορετικό από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό περιπλέκει την δυνατότητα εγκατάστασης, ε, την ομοιογενή διαχείριση. Τι μπορείτε να κάνετε ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αποκλίσεις, τις διαφορές και να μπορεί να υπάρχει ελευθερία εγκατάστασης. Ναι, εάν κάτι τέτοιο έχει νόημα θα το κοιτάξω. Πάντως, εξ όσων θυμάμαι, κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις ήταν συνήθως εξαιρετικά τοπικού χαρακτήρα και μπορούσαν να συμβάλλουν στη συνοχή μιας ε, κοινωνίας. Δηλαδή σε χώρες όπου κάποιοι ε, ε, κατάφεραν έτσι να αισθανθούν λιγότερο εγκαταλελειμμένοι. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο να εργαστούμε από αυτά αυτή τη στιγμή, όμως γιατί όχι. Έχουμε συζητήσει να δημιουργήσουμε ιδρύματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα, ώστε να μπορούν να γίνουν και δωρεές διασυνοριακές ο κύριο Μπέρ νομίζω έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ε, η κυρία Νίκολα Μπέρ έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρε τέτοιε δραστηριότητε ε, διασυνοριακώ. Προσανατολισμού έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, Ένα επίτροπο θεωρώ ότι πρέπει να συνεργάζεται με τι υπηρεσίε του και να δίνει κάποιε επιταγέ, κάποιε κατευθύνσει. Σα διαβεβαιώ ότι οι ενδείξει και οι κατευθύνσει θα υπάρξουν σαφώ δυναμικές από την πλευρά μου. Invest EU, νομοθετική διάσταση, επιχειρήσεις, όλα αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Επόμενος ο κύριος Τζούλο από τους μη εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ υποψήφια Επίτροπε. Ήθελα να επαναλάβω κάποια από τα πράγματα που επαναλάβατε σήμερα επανειλημμένως. Έναν από τους στόχους δηλαδή να έχουμε από άποψη κλιματικών αλλαγών στο 2050 μια ήπειρο ουδέτερη, διαχειριζόμενη τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάση των εμπειριών της προηγούμενης θητείας και όσων συζητήσαμε με την Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα πρέπει, πρέπει να υπάρξει μια μετάβαση που να έχει ως κέντρο της την κυκλική οικονομία, κοιτάζοντας και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων αυτή τη στιγμή είναι προφανές σε όλους ότι οι ηλεκτρικές μηχανές, τα οχήματα έχουν πολύ μικρότερο κύκλο ζωής από το παρελθόν. Και δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι βιώσιμο ούτε από την οικονομική ούτε από την ηθική σκοπιά. Πώ τη βλέπετε λοιπόν αυτή τη μετάβαση προ μια οικονομία που επιτρέπει την διάρκεια, μεγαλύτερη διάρκεια ζωή των προϊόντων, την δυνατότητα επισκευή του, πώς θα γίνεται να καλυφθούν αυτά τα κενά. Ευχαριστούμε κύριε Τσούλο, ε, κυρία Γκουλάν. Ευχαριστώ, χαίρομαι που ακούω λίγο Ιταλικά, γιατί δεν είναι και τόσοι πολλοί ευρωβουλευτέ από την Ιταλία που πήραν σήμερα το λόγο. Για το θέμα αυτό της διάρκεια ζωή των προϊόντων και την εφορία του. Έχουμε πραγματικά φιλοδοξία να κάνουμε κάτι. Και νομίζω ότι και πάλι είναι πολύ σημαντικό και για τους πολίτες. Ε, εάν αποδείξουμε ότι κάνουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι συγκεκριμένο, όταν πάνε να κάνουν τα ψώνια τους, όταν πάνε κάτι να αγοράσουν ε, κάτι, και βλέπουν μέσα σε μια πενταετία υπάρχουν λιγότερα πλαστικά και υπάρχει μια διαφορά στην καθημερινότητά του. Προτεραιότητα λοιπόν αναμφίβολα. Αλλά και εδώ θα ήθελα να παραμείνω κάπω συγκρατημένη, διότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν δυνατότητε και ευκαιρίε για ένα μεγάλο κομμάτι τη οικονομία για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Όμω δεν πρόκειται για κάτι που είναι εύκολο να αναλάβει κανεί δράση. Για τα τρόφιμα, για τα κλωστοεφαντουργικά και τα ενδύματα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε ξεκινήσει, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Και στα Ιταλικά νομίζω λέγεται, λέτε συχνά ε, προγραμματισμένη λήξη ζωής. Εδώ είπαμε να κάνουμε κάποιε δοκιμέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 για να δούμε αν αυτό συμβαίνει όντω ή όχι. Αλλά πρέπει να πάμε και παραπέρα τι γίνεται τώρα με κάποια προϊόντα που δεν πολλούνται. Να, να καταστρέφουμε, να τα αποσυναρμολογούμε. Όταν μιλήσαμε για την καταπολέμηση, όταν μάλλον ασχολήθηκα με την καταπολέμηση τη φτώχεια, είχα πάει στην Ιταλία και συζήτησα σχετικά με ενώσει. Ε, ενώσει που λέγανε ότι δεν μπορούμε πλέον να σπαταλάμε, να πετάμε στα σκουπίδια τόσα τρόφιμα. Και υπάρχει και το θέμα τη ενημέρωση του καταναλωτή για τη διάρκεια ζωή των προϊόντων του. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει και να βελτιωθεί. Αλλά είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και πρέπει να είμαστε και κάπω συγκρατημένοι. Διότι πάνε μακριά. Σκοπό πάντω είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Να αλλάξουν. Νομίζω ότι σταματάμε τα τελικά. Κουράστηκα, ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να παρακολουθώ και τι σημειώσει μου στα γαλλικά ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρα. Επερώτηση κύριε Τζούλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πίτροπε. Ε, εκτιμώ την προθυμία σας και αυτή τη διάθεση να κοιτάξετε πώς θα περιοριστούν οι διάφορες σπατάλες. Ένα από τα αποτελέσματα που αποσπάσαμε στο Κοινοβούλιο συζητώντας για το θέμα αυτό είναι ότι το να προωθήσουμε τη διάρκεια ζωή σημαίνει ότι προωθούμε και ένα νέο τρόπο ζωή, μοντέλο ζωή. Δηλαδή να εργάζεται κανεί σε τοπικό επίπεδο, όχι αποκεντρωμένα ε, και ότι δίνουμε νέα ζωή στην Ήπεθρο. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να το θέσουν αυτό στόχο και μπορούν έτσι να αποσπάσουν αποτελέσματα και σε ε, λογικό χρονικό διάστημα. Θα μπορούσαμε να υποχρεώνουμε ή να προβλέψουμε αυστηρέ προποθέσει για προϊόντα και μετά τα ανταλλακτικά να ε, προσφέρονται χωρίς τεράστιες ε, προσαυξήσεις και διαφορές τιμών ελπίζω λοιπόν αυτό να προχωρήσει και εσείς να γίνετε αυτοί που θα προωθήσει ακριβώς προσωπικά αυτό το στόχο. Σας ευχαριστούμε κύριε Τζούλο. Κύριε Γκουλάρ. Υπάρχει κάθε διάθεση, αλλά πρέπει να υποχρεώσουμε όπως λέτε, έχετε δίκιο. Πρέπει όμως και να εκπαιδεύσουμε. Ε, αυτά πάνε μαζί. Δεν μπορεί κανείς απλώς να πιθαναγκάζει. Πρέπει να αφήσουμε και λίγο χρόνο στις επιχειρήσεις για να κάνουν αυτήν την ε, μεταβολή, αυτήν την αλλαγή. Συζητήσαμε πάντως και προηγουμένω το παρελθόν μαζί μας, λόγω χάρη, μεταξύ μα λόγω χάρη για τα απόβλητα. Και συζητήσαμε για τα απόβλητα, ε, τον τι είχε καταναλωθεί και τα απλά απόβλητα. Όπως λέτε, Έπρεπε να αλλάξει τελείω όλη η αλυσίδα παραγωγή και να ε, σχεδιάζουμε τα προϊόντα με έναν τρόπο τελείω διαφορετικό για να φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή να περιοριστεί το μερίδιο, το τεμάχιο αυτό των ε, αποβλήτων. Είναι κρίμα να πετιώνται όντω τα τρόφιμα και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταναλώνουμε τα προϊόντα αυτά ακριβώς, αλλά με τρόπο εντελώς διαφορετικό. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Πέτρα Κούμπουλα Νάτρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κυρία Γκολάρ, βασιζόμαστε στη δική σας δουλειά όσον αφορά την ψηφιοποίηση. Χρειαζόμαστε γρήγορε συνδέσει για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και ανάπτυξη στην Ευρώπη και να καταπολεμήσουμε την ε, αλλαγή του κλίματο. Χρειαζόμαστε λοιπόν καινοτόμες τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ελπίζω να θεωρείτε ότι χρειάζονται ρύθμιση οι ψηφιακές ε, οικονομίες. Ε, πρέπει να διασφαλίσουμε τον ιδιωτικό βίο και να ε, προστατεύσουμε τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Οι αγορές δεν μπορούν να το κάνουν αυτά μόνα τους. Δύο ερωτήσεις. Είσαστε διατεθειμένοι χωρίς επιφύλαξη να προωθήσετε τις ε, γρήγορες ε, συνδέσεις ε, και, την, και το 5G για όλους. Και δεύτερη ερώτηση, θα προτείνετε νέα νομοθεσία για το roaming, για την περιαγωγή και τις διεθνείς, και τις διεθνείς εκκλήσεις. Νομίζω ότι όλα θα έχουν ένα τέλος σε λίγα χρόνια. Ναι, απάντησε στην όχι. Σε ό,τι αφορά τη γενιά 5G, δεν υπάρχει καμία συζήτηση πλέον. Θα παρασταθούμε όσο γίνεται στις χώρες μέλη για να προσαρμοστούν σε εξελίξεις που είναι πολύ σημαντικές για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με σεβασμό φυσικά όλων των κανόνων για τη δημόσια υγεία. Θα γίνει σταδιακή αξιολόγηση. Πάντως, το ψηφιακό χάσμα είναι αισθητό γιατί έχουμε μερικές απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν ευρυζωνικότητα. Και αυτό συν... επιτείνει τον αποκλεισμό τους. Το 2019 μόνο 5% των αγροτικών νοικοκυριών είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ ε, και 60% ευρυζωνική. Οπότε ε, βλέπετε ότι είναι δύσκολο και πρέπει να καλύψουμε αυτό το ψηφιακό κενό. Το 60% συγγνώμη δεν είχαν ευρυζωνική. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα για τις επενδύσεις στον τομέα αυτό, το ψηφιακό και φυσικά να λειτουργήσει και ο ανταγωνισμός για την ε, κατανομή του ραδιοφάσματος και το καθεξής. 3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, αφιερώνοντας το πρόγραμμα στην Ευρώπη, το πρόγραμμα για τη διασύνδεση της Ευρώπη και να συνδέσουμε τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλους τους διάβλους διασυνδεσιμότητας ή διασύνδεσης. Επίσης, είχαμε μια πρωτοβουλία που βοηθούσε τους Δήμους να προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi με συγκεκριμένη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση των διεθνών κλήσεων, όσα έγιναν για την περιεγωγή στην Ευρώπη ε, έγιναν ε, δεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό και ήταν πολλοί οι πολίτες που υποφελήθηκαν, φοιτητέ, νοικοκυριά και ούτω καθεξής. Θα δούμε πώς ε, θα συνεχιστεί η κατάσταση και θα λάβουμε τα μέτρα για να πολλαπλασιάσουμε τα ωφέλη του roaming. Πάντως πρέπει να γίνει πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για να δούμε τι μέτρα θα προτείνουμε στο μέλλον. κυρία Κούπουλα Νάτρη έχει επερώτηση. Η πολιτική προσήλωση φυσικά είναι το πιο σημαντικό στη φάση αυτή. Κυρία Επίτροπε, ε, τρεις γενικέ διευθύνσει θα έχετε από την αρμοδιότητά σας, ε, την εσωτερική αγορά, την βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσει, ε, ψηφιοποίηση. Ζώμαστε ψηφιοποίηση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Χάνουμε στους πιο σημαντικούς τομείς. Ε, διάβασα ότι λιγότερο από το 3% τα 100 των καινοτομιών ε, στον τομέα αυτών ε, δημιουργείται από Ευρωπαίους. Κάτι τέτοιο όμως θα ήταν καλό και για τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Πολύ συγκεκριμένα, πόσες μέρες την εβδομάδα, 5 ή 7, ε, θα χρησιμοποιείτε ε, για, θα αφιερώνεται στην Γενική Διεύθυνση Connect, στην Γενική Διεύθυνση της Εσωτερικής Αγοράς ε, και στην Γενική Διεύθυνση για, για το διάστημα. Ναι, δύσκολη ερώτηση, γιατί Μπορεί να σας φαίνεται τεράστιο απέραντο το χαρτοφυλάκιό μου, γιατί έχουμε δύο γενικές διευθύνσεις που ήδη υπάρχουν και μία ε, που είναι στα σπάργανα. Ε, ουσιαστικά θα είναι τρει δηλαδή. Και όντω, στα ψηφιακά ζητήματα διατρέχουμε τον κίνδυνο στην Ευρώπη να μείνουμε πίσω σχέση με άλλε χώρε. Και σίγουρα η ψηφιοποίηση θα είναι κορυφαία μας δραστηριότητα. Τώρα τι χρόνο θα αφιερώνω στην Γενική Διεύθυνση Connect, να σας πω, αυτό είναι πολύ αφηρημένο. Πάντως, η ακράδαντη πεποίθησή μου είναι ότι η ψηφιοποίηση των οικονομιών μας θα, την, θα πρέπει να ωφελήσει τη βιομηχανία, να λάβει υπόψη τον πολιτισμό, να συνδυαστεί με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, γιατί είναι αδιανόητο ε, να μην γίνουν πιο φιλοπεριβαλλοντικές οι επιχειρήσεις και να διαχωρίσουμε αυτή την προσπάθεια από, από την ψηφιοποίηση. Πάντως είναι πολύ αφηρημένο όλα αυτά. Δεν μπορώ να σας πω πόσες ώρες θα θυρώνω στη μία γενική διεύθυνση και πόσες στην άλλη. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι θα εργαστώ σκληρά, θα με συνέχεια στις Βρυξέλλες και αν μην Νομίζω ότι αν σα πω πόσε ώρε αφιέρωσα την τελευταία εβδομάδα στι διάφορε οδηγίε, μην το πείτε σε αυτού που ασχολούνται με την επιβολή νόμου. Πραγματικά ε, κάναμε σκόνη την οδηγία για το χρόνο, για το ωράριο εργασία. Κυρία Βαλεάν, αναλαμβάνει την Προεδρία. Συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ο κύριος Ιβαν Στέφανετς στην Επιτροπή ΙΜΚΟ από το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Οριστήσα Επίτροπε, εδώ είμαι. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όσον αφορά τις αρχές που αφορούν ε, την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων ανθρώπων και προϊόντων, διότι οι αρχές αυτές δεν λειτουργούν πάντα πολύ καλά στην πράξη. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας αυτοαπασχολούμενος αρχιτέκτονας από το Λουξεμβούργο θέλει να πάει στη Γαλλία. Αυτό μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα, διότι υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, αλλά Εάν το ίδιο πρόσωπο θέλει να φέρει και κάποιον για να τον απασχολήσει, τότε είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Διότι πριν την πρόσληψή του θα πρέπει να γίνει η απόσπαση και υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται Κάτι που καθιστά ε, αυτό σχεδόν αδύνατο. Ουσιαστικά λοιπόν η ελεύθερη κυκλοφορία δεν λειτουργεί πολύ καλά. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοια γραφειοκρατικά εμπόδια ώστε η εσωτερική αγορά να λειτουργεί στην πράξη. Κυρία Γκουλάρ, ευχαριστώ κύριε Στέφανετς που δώσατε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με επαγγέλματα. Γιατί Βλέποντας τις στατιστικές για τις παραβιάσεις, συνειδητοποιούμε ότι ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται η ελευθερία εγκατάστασης για τα ρυθμισμένα επαγγέλματα. Φυσικά δεν είναι εύκολα αυτά τα ζητήματα γιατί οι χώρες έχουν τις παραδόσεις τους. Αυτό είναι θετικό βέβαια. Και όταν έχουν να κάνουν με κάποιον επαγγελματία θέλουν να είναι καλά εκπαιδευμένος, να έχει τις δεξιότητες όταν προσλαμβάνει κάποιος αρχιτέκτονα θέλει να είναι σίγουρος ότι το σπίτι του θα έχει ένα θεμέλια. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα υπερβούμε αυτό το σκόπελο. Πάντως, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εφαρμόζει συστηματικά τις οδηγίες για τα επαγγελματικά προσόντα και τις επαγγελματικές δεξιότητες. Είναι σημαντικό, λοιπόν, ε, να φέρουμε στο επίκεντρο ένα τομέα ε, και να κάνουμε πράξη την ελεύθερη διακίνηση. Γιατί μιλήσαμε για τέσσερι ελευθερίε και θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι τέσσερι. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει με τι διαδικασίε επιπαραβάση, μπορεί να γίνει με το διάλογο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μερικέ φορέ ε, υπάρχουν κάποια συντεχνιακά συμφέροντα. Κάποια επαγγέλματα ε, είναι κλειστά και θέλουν να παραμείνουν κλειστά, να κρατήσουν τα προνομιά του. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν την ισορροπία μεταξύ τη ε, εύλογη και θεμητής προστασίας που, συνοδεύεται, που συνοδεύει το πτυχίο και από, μεταξύ αυτού και της υπερβολικής προστασίας. Επίσης, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη μερικά πράγματα και ίσως με βγάζετε λίγο εκτός του χαρτοφυλακίου Αυτό είναι θέμα απασχόλησης και του Επιτρόπου Νικολά Σμιτ. Και σίγουρα θα εγγύψει αυτά τα θέματα με το που θα αναλάβει τα καθήκοντά του για να προσφέρει λύσεις σε όλους τους επαγγελματίες που προβληματίζονται. Επερώτησα από τον κύριο Στέφανετς. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Η παρατήρηση που έκανα έχει να κάνει και με τον καθημερινό αγώνα κατά της γραφειοκρατίας και για την εξάλληψη των εμποδίων. Και πιο προβληματικός είναι ο τομέας των υπηρεσιών. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σας προσέγγιση. Πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε στον τομέα των υπηρεσιών. Και από νομοθετικής πλευράς πρέπει να προχωρήσουμε. Θα ξανανοίξετε την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ή θα προτιμήσετε άλλη μέθοδο. Αυτό που δείχνει και η συζήτηση σήμερα είναι ότι ανάλογα με το ποιο θέτει την ερώτηση από ποια χώρα προέρχεται, τη προσδίδει διαφορετικό νόημα. Η κυρία Γκέπχαρτ είπε πριν από λίγο ότι θα πρέπει να ξανανοίξουμε συζητήσει ε, που χωρίς λόγο θα προκαλέσουν αντιδράσεις, αλλά εσείς ζητάτε ε, το αντίθετο. Βέβαια, δεν μπορώ να αρκεστώ στην προσωπική μου γνώμη, γιατί η προσωπική μου γνώμη όταν κανεί είναι μέλο ενό συλλογικού οργάνου δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να σεβαστώ και τις γνώμες των συναδέλφων επιτρόπων και κυρίως το αρμόδιο για την απασχόληση. Πάντως το θέμα άπτεται και της ενιαίας αγοράς, οπότε αναγκαστικά θα ασχοληθώ και εγώ με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και γνωρίζετε πως μερικές φορές η κοινή γνώμη ε, κατηγορεί μερικούς, ε, κινδυνολογεί μερικές φορές, ε, μιλά για απειλές, ε, και χειρίζεται πολύ αρνητικά αυτά τα ζητήματα. Ε, σίγουρα θα πρέπει να βρούμε λύσεις χωρίς να υπονομεύουμε τα κοινωνικά δικαιώματα που φυσικά είναι προσφυλή στον κόσμο και να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Ο κύριος Μανουέλ Μομπάχ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκουλάρ, χαίρετε. Συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις των ε, πολυάριθμων συναδέλφων που μίλησαν για τις οντολογικές δυσκολίες που μας θέτει η υποψηφιότητά σας. Όμως για τη μηχανική πολιτική, πέραν όλων αυτών, που αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου σας, θα Μα πείτε φαντάζομαι κι εσεί ότι είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία σήμερα ειδικά γιατί χρειαζόμαστε μια οικολογική μετάβαση. Η πραγματικότητα είναι σκληρή σήμερα. Η Ευρώπη έχει χάσει εκατομμύρια θέσει απασχόληση στι βιομηχανίε και τι εταιρείε τη τα τελευταία χρόνια και είναι πολλοί οι τομεί που είναι απαραίτητοι στην οικολογική αυτή μετάβαση. Απειλούνται όπω η χαλιβουργία, η μεταλλουργία, οι βιομηχανικέ παραγωγέ όπω η Alstromin, σαν Κομπάν στη Γαλλία, ε, είτε πολλούνται τα εργοστάσια του, είτε υπάρχει περίπτωση περίπτωση να Εδώ στι απαντήσει σα στο ερωτηματολόγιο, λέτε ότι τα θέματα αυτά τη βιομηχανική στρατηγική σα απασχολούν ιδιαίτερα. Πέραν όμω των δηλώσεων και των λόγων Ποιες είναι οι απτές σας δεσμεύσεις, θα προβλέψετε οικολογικούς φόρους υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κάνετε πιο ευέλικτους τους κανόνες για τις κρατικές βοήθειες, ώστε να μπορούν να προβάλλουν ε, ανεξάρτητες εθνικές στρατηγικές τόνωσης των ε, βιομηχανιών τους και να ε, διακόψετε τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που μας οδηγούν σε πλήρη απελευθέρωση, τονώνοντας την βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλάρ. Κοιτάξτε κύριε Βουλευτά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιομηχανική πολιτική θα είναι μια από τι προτεραιότητε και αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν με εμπιστευτείτε όλο ιδιαίτερω εμού τη ιδείας. Και γιατί. Διότι αν θέλουμε από τη μια πρασίνισμα και από την άλλη ψηφιοποίηση, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρί βιομηχανία. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τι θέσει απασχόληση στην Ευρώπη, Βεβαίω, ε, πολλά θα πάνε στη Γεωργία, πολλά στην ε, ε, σε άλλους χωρούς, αλλά υπάρχουν, παρά, υπάρχει παράδοση και ιστορία στην Ευρώπη. Πολλοί είναι τομείς που πρέπει να διαφυλαχθούν. Ε, φόροι, ε, το είπε η κυρία Φοντερ Λάιεν, το έχουμε συζητήσει από καιρό. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μελετηθεί, ε, παρόλο που επί χρόνια ήταν ταμπού. Και πρέπει να δούμε ξανά την παραγωγή, γιατί έχουμε αλυσίδα παραγωγής με... Ε, μια εξισορρόπηση εισαγωγών-εισαγωγών στου δασμού που πολλέ φορέ δεν συμφέρει την Ευρώπη. Το έχουν δει και οι Αμερικανοί και βλέπουν δεν του ε, συμφέρει. Δεν έχω λοιπόν εδώ κανένα ταμπού, αλλά πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Να δούμε τι είναι συμβατό με του κανόνε του ΠΟΕ. Και να σκεφτούμε, οι κανόνε του ΠΟΕ θα πρέπει να ε, δυσλειτουργούν και να μην έχουν σωστή εφαρμογή. Θα το πρέπει να το δούμε. Σε ό,τι αφορά τι κρατικέ βοήθειε, πιστεύω ότι υπάρχει ένα τρόπο να βρούμε λύση Σημαντικό τρόπο, τον οποίο τον ανέφερα και προηγουμένως στα λεγόμενά μου. Πρέπει να έχουμε τέτοιου ε, τομεί όπου να μπορούμε να ε, στείλουμε, να δώσουμε δημόσιο χρήμα. Το είπα, η διασυνδεμένη υγεία, ε, αυτοκινητοβιομηχανία και το καθεξής. Αλλά εδώ πρέπει να διασυνδέσουμε τους δημόσιου πόρους ενθαρρύνοντας τις εταιρικές σχέσει με τον ιδιωτικό τομέα θα γίνει τώρα αυτό αλλάζοντα το σύστημα κρατικών βοηθειών υπό την έννοια ότι θα επιτρέψουμε στι κρατικέ δυνάμει σε όλε τι περιπτώσει, για όλα τα θέματα, για οποιαδήποτε επιχείρηση. Πιστεύω ότι θα ήταν υπερβολικό. Όμω οι εταιρείε μα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρίσκονται σε παγκόσμιο ανταγωνισμό με, χω... με χώρε που πολλέ φορέ στηρίζουν, είτε με μεντικά προγράμματα είτε με άλλα, τι επιχειρήσει του απολύτω. Το δώμα τώρα. Ε, εγώ θα ε, περιοριστώ να κάνω τη δουλειά μου και τίποτα περαιτέρω. Ευχαριστώ για την απάντησή σας, αλλά μου φαίνεται λίγο φλού, λίγο ασαφής. Δεν μπορείτε απλώ να μα λέτε όπω πολλοί άλλοι επιτροπή. Θα το συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε στο μέλλον. Σήμερα θέλουμε να ξέρουμε τι θα κάνετε, όχι σε πέντε χρόνια, όταν θα τα έχετε συζητήσει. Βεβαίω ε, είναι θέμα, δεν είναι, δεν θρησκευτική, θρησκοληψία το όλο θέμα. Και βεβαίω το δόγμα είναι θέμα θρησκεία, όμω στην Ευρώπη δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα γιατί η, η, ιδέα της, των ελεύθερων συναλλαγών και τη απελευθέρωση είναι ο μόνο μπουσουλά. Μα οδηγεί σε καταστροφή τη βιομηχανία μα, του βιομηχανικού ιστού, του περιβάλλοντο και των κοινωνικών σχέσεων. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθείτε ότι εφ' θα Σχεδιάστε και θα έχουμε πλέον μια στρατηγική για να σχεδιάσουμε τη βιομηχανία όπω θέλουμε και να αναπτυχθεί στην Ευρώπη. Να προστατεύσουμε επιτέλου την τεχνογνωσία, τα στατικά μα συμφέροντα και τα συμφέροντα των εργαζομένων μα έναντι όσων σε διεθνέ επίπεδο δεν ε, λαμβάνουν την ίδια προσοχή για τα μεγάλα αυτά κοινωνικά και οικολογικά θέματα. Κύριε Γκουλάρ. Συμφωνώ με αυτό που μόλις είπατε. Και όντω η στρατηγική που εγκρίθηκε για την Κίνα, χωρί να θέλω να στιγματίσω καμιά χώρα ή να την, να την κάνω δεκτυλοδεκτούμενη. αλλά αυτό που έχουμε συζητήσει δείχνει ότι υπάρχει μια συνειδητοποίηση που έλειπε πριν από δύο-τρία χρόνια αντίληψη αυτή ότι έχουμε ανταγωνιστές που είναι όμως και τέρι. Το είδα στην ε, διάθεση των, ε, από την Τράπεζα της Γαλλίας, στη διάθεση των Κινέζων, να είναι φίλοι και σύμμαχοι στα θέματα του κλίματος. Δεν είναι τα πράγματα τόσο μονόδρομα. Ούτε όμως πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις απέναντι σε τέτοιες χώρες. Δική μας δουλειά, όλων μας, είναι να βρούμε τον ευρωπαϊκό δρόμο δεν μπορούμε να ζήσουμε σε ένα κόσμο διαφορετικό από αυτόν τον οποίο ζούμε. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε το πεντάγωνο, το πεντάγωνο επιδοτεί επιχειρήσει ε, αμερικανικέ. Οι Κινέζοι από την πλευρά του κάνουν κάτι αντίστοιχο. Εμεί όμω έχουμε ως πλεονέκτημα το να παραμείνουμε ανοιχτοί. Όχι αφοπλισμένοι, όχι, όχι. Βλέπω το body language σα και τη γλώσσα του σώματο και τι εκφράσει σα. Όχι θα ψάξουμε όλες τις ε, κατευθύνσεις. Θα είμαστε ανοιχτόμυαλοι, αλλά όχι ε, ανοιχτοί σε όλα. Ευχαριστούμε κυρία Κάμερεβερτ. Από την Επιτροπή Πολιτισμού, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση της συναδέλφου Φερχάιεν. Γιατί η απάντησή σας, ε, κύριε Γκουλάρ, δεν με έπεισε συνολικά στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, προσφορές και μεγάλη ζήτηση για πακέτα με ειδήσει μέχρι και για σινεμά. Εδώ λοιπόν ξέρουμε ότι υπάρχει μια συναρπαστική πολιτιστική διάσταση, την οποία βλέπουμε και στην Επιτροπή μας. Στην απάντησή σας, όπτικα, ακουστικά, μέσα, δεν διαβάσουμε πουθενά. Ε, και ε, είναι θέμα ευρωπαϊκού δικαίου. Πρέπει και εκεί κάτι να προβλεφθεί. Τα, κρα... τα κράτη-μέλη μόνα του δεν μπορούν πλέον να τα αναλάβουν όλα μόνα του. Είναι προφανέ. Οπότε, ω επίτροπο, έχετε καμιά ιδέα για το τι κατεύθυνση θα πρέπει να πάρουν τα πράγματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πώ σκέφτεστε στο πλαίσιο τη πράξη για, την... Ε, για τι ψηφιακέ υπηρεσίε να κάνετε κάτι και για τα οπτικοακουστικά και αυτού που πραγματικά ξεχωρίζουν να του υποστηρίξετε περαιτέρω ώστε τα, ε, τηλεοπτικά προγράμματα που αξίζουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ, κυρία κάμερα. Σα ευχαριστώ που επιτρέπετε να επανέλθω στο θέμα αυτό. Δεν, δεν ήθελα να δώσω την εντύπωση, λαντασμένα, ότι δεν με ενδιαφέρει ο πολιτισμό αυτό καθεαυτό. Δεν αληθεύει και ακόμη περισσότερο η πολιτιστική ποικιλομορφία όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ σε αυτή την αίθουσα, τελικά πρέπει να αναρωτηθούμε τι είναι η Ευρώπη. Είναι τόση πολλή ποικιλομορφία σε ένα τόσο μικρό χώρο. Είναι φανταστικό να έχουμε αυτή τη δημιουργία η οποία εμπλουτίζεται από τι επιρροέ των ΕΝ και των ΔΕ σε ένα χώρο τόσο μικρό και να υπάρχει και αμοιβαία αλληλεποστήριξη. Άρα η προβολή του πολιτισμού και τη παιδεία είμαι τελευταία που δεν θα το, δεν θα το ήθελα αυτό. Ε, Στι απαντήσει τη ερωτήσει εδώ στην Ακροασία έχει κανεί πολύ λίγο χρόνο στη διαδικασία του. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Τώρα, ο χώρο των απτικοακουστικών πραγματικά ε, περνάει από μια ψηφιακή μεταμόρφωση όπω και άλλοι κλάδοι. Αλλά υπάρχει και το θέμα των πλατφορμών για εδώ που είναι πολύ σημαντικό, τη μετάδοση, τη δίκαιη αμοιβή όσων έχουν τα δικαιώματα πνευματική υπηρεσία, τη προσφορά και τη ζήτηση. Πολύ περίπλοκα συστήματα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά δηλαδή, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μειωθεί η προάσπιση τη ποικιλομορφία. Όσο για το Creative Europe, το πρόγραμμα για τα μέσα, νομίζω, είναι περίπου το μισό του προπολογισμού αυτού του προγράμματο. Νομίζω ότι έχει πετύχει. Οι, οι εταιρείε των διαφόρων κλάδων συνεργάζονται υπάρχει μεγάλη παραγωγή ταινιών και όταν πηγαίνω στον κινηματογράφο πραγματικά μου κάνει εντύπωση που βλέπουμε ότι ο πολιτισμός πλέον δεν πηγαίνει μόνο στις πρωτεύουσε, αλλά και στις μικρότερες πόλεις της επαρχίας. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτός ο ανταγωνισμός να διατηρηθεί με την υποστήριξη που είπαμε και για κάποιες ε, τηλεοπτικές σειρέ. Άρα οι ταινίε ε, που έχουν υποστηριχθεί πολλές φορές έχουν κερδίσει και διεθνή βραβεία και σε καμία περίπτωση δεν τα πειράζουμε αυτά. Τώρα πώς μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα για την πτυχή Creative Europe σε συνεργασία με τα μέσα. Είναι όντω αποσυνδεδεμένα αυτά τα δύο. Η γενική διεύθυνση με την οποία ασχολούμαι εγώ και αυτή τη Μαρία Γκάμπριελ. Όμω θα κοιτάξουμε να συνεργαστούμε. Η εμπειρία τη θα μου είναι πολύτιμη και ξέρω ότι έχει δουλέψει ήδη μαζί σα για τα θέματα αυτά. Οπότε πιστεύω ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να πάμε και μακρύτερα. Επερώτηση. Κυρία Καμερέβερτ. Ευχαριστώ για την απάντηση. Όμως, Τελικά δεν απαντήσατε πραγματικά στην ερώτησή μου. Εγώ ρώτησα ποια συγκεκριμένα μέτρα, τι συγκεκριμένε ιδέε έχετε για τον τομέα των οπτικοακουστικών ω παράγοντα πρόθεση του πολιτισμού και τη παιδεία στην Ευρώπη. Πώ θα τον ενδυναμώσετε, Μπορείτε να μα πείτε ένα αντίβαρο που θα βρείτε εδώ σε σχέση με του Αμερικανού παραγωγού στον τομέα αυτό. Δεν άκουσα τίποτα σχετικό. Θα ήθελα κάτι λίγο πιο απτό, λίγο πιο συγκεκριμένο. Μπορείτε να γίνετε συγκεκριμένοι. Πολλέ φορέ είπατε ότι θα τα συζητήσετε, θα τα πείτε, θα τα βρείτε. Ιδέε όμω θέλουμε, κάτι συγκεκριμένο. Σε ποια κατεύθυνση θα πάτε, Κυρία Γκουλάρ, ευχαριστώ. Για να σας τα πω, ίσως λίγο πιο ευθέως. Προφανώ η διαφύλαξη τη ποικιλομορφία και των μικρών παραγωγών σε σχέση με του κολοσσού που έρχονται από άλλε περιοχέ του κόσμου και έχουν πολύ χρήμα στη διάθεσή του, επί τη αρχή είναι κάτι το οποίο με βρίσκει απολύτω σύμφωνο μαζί σα. Οπωσδήποτε θα δώσουμε αγώνα για την ποικιλομορφία, αλλά το δείτε και μόνοι σα. Ε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εγώ παίρνω την πραγματικότητα ως έχει και την Ευρώπη ως έχει. Σε τομείς που ως τώρα ε, δεν είχα ακουμπήσει στη δουλειά μου. Ε, δεν θα πω εγώ ότι τώρα επειδή ήρθα εγώ θα πάψουν οι μεγάλες πλατφόρμες να ε, συνεχίζουν την προέλασή τους. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά την κατεύθυνση θέλουμε να την ακολουθήσουμε. Τώρα το πώς θα φτάσουμε ως εκεί. Πολύ ειλικρινώς δεν θέλω να σας φανώ υπεροπτική και να σας πω ότι τη λύση την έχω. Έχω την τέλεια συνταγή και θα το καταφέρω. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Ε, thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Σπάνεντακ. Συγγνώμη, η κυρία διορθώνει η πρόεδρο. Oh, wow. ε, δεν, σα έχω γνωρίσει ακόμα. Η κυρία Κιμ Φαν Σπάρεντακ. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει σα Εδώ κάθομαι. Η εκλεγήσα πρόεδρος ε, δεσμεύτηκε να ε, μειώσει τις ε, εκπομπές στη βιομηχανία, το να έχουμε μια ουδέτερη ε, ως προς το διοξείδιο του άνθρακα περιβάλλον θα είναι μεγάλη πρόκληση. Πώς ε, σκοπεύετε να δώσετε αρκετά κίνητρα για να έχουμε πιο πράσινες δημόσιες συμβάσεις στην εσωτερική αγορά. Θα αναθεωρήσετε την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Προβλέπετε νέα μέτρα για οι φόρες ε, αλυσίδες προμήθειας και θα συμπεριλάβετε τα σχετικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσει, Κυρία Κουλάρ. Ναι, αυτή την άγουσα θα ακολουθήσουμε με αποφασιστικότητα. Και το μήνυμα που θα ήθελα να διαβάσω σήμερα είναι ότι αν με εγκρίνετε, εννοείται, αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, η Επιτροπή θα επιταχύνει το πρασίνισμα με βάση τα μέσα που έχουμε. Οι δημόσιες συμβάσεις είναι 14% των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε θα υπάρξει μόχλευση. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Επίσης, όταν έχουμε ένα τοπικό αιρετό, ε, αυτό που κάνει την επιλογή, φυσικά τον ενδιαφέρει και η τιμή που θα πληρώσει. Και μερικές φορές ε, υπόκεινται οι αιρετοί στον έλεγχο των ε, ψηφοφόρων, γιατί χειρίζονται δημόσια κονδύλια, οπότε το κόστος είναι σημαντικό. Θα γίνει μια φυσικά αλλαγή της ε, νοοτροπίας, χρειάζεται, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το διευκολύνουμε. Επίσης μιλήσαμε για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και για να σημειώσουμε πρόοδο δεν θα πρέπει να πρασινίσουμε μόνο τις διαδικασίες, θα πρέπει ένα ολόκληρο τμήμα της κοινωνίας που εργάζεται διαφορετικά κοινωνικά, φιλοπεριβαλλοντικά, ε, λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση των φίλων με αλλαγή στις διαπροσωπικές σχέσεις. Όλες αυτές τις αλλαγές θέλουμε. Και γι' αυτό οι, αποφάση αποφάσεις για τις δημόσιες συμβάσεις είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Επίσης, τα κοινωνικά κριτήρια υπάρχουν ήδη, περιβαλλοντικά κριτήρια. Ε, και ήδη οι φορείς για τη χάραξη πολιτικής μπορούν να τα εφαρμόσουν. Επίσης, ε, θέλουμε κάποιο είδους κατάρτιση για τους ηθήνοντες πολιτικής. Αυτό θα ήταν χρήσιμο για να προωθήσουμε αυτή την ιδέα. Και σίγουρα αυτό το εργαλείο θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Επερώτηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά τους σπόρους και την ανάγκη να ε, περιορίσουμε το ε, οικολογικό μας αποτύπωμα, τι μέτρα προτείνετε για την οικονομία της εσωτερικής αγοράς. Δεσμεύεστε να θέσετε στόχο για την ε, αποδοτικότητα των πόρων ως μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η κυρία Γουλάρ; Ήδη προβλέπονται κονδύλια στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και είμαι σε δύσκολη θέση, το είπαμε προηγουμένως και στον συνάδελφο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το ύψος των κονδύλιων στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Υπάρχει ένα οικονομικό σκέλος για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή νοτροπίας υπέρ της κυκλικής οικονομίας. Και φτάνουμε πραγματικά στο σημείο καμπής, ε, που θα έχουμε και επικερδείς επιχειρήσεις που θα είναι ταυτόχρονα και αλληλέγγυες. Δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο ε, κάποιους που θα υλοποιούν το στόχο, αλλά θα τον υλοποιούν με κερδοφόρο τρόπο. Επίσης, ε, για την ε, διαχείριση των αποβλήτων, θα πρέπει και η ανακύκλωση να γίνει ε, επικερδής. Και ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα αυτά είναι από τη δική σας πολιτική οικογένεια, είναι πολύ δυναμικός και ενθουσιασμένο, είναι 28 χρόνο μόλι πολύ νέο. και νομίζω ότι θα μας φέρει τη σκοπιά των προσδοκιών των νέων γενιών για τα θέματα του περιβάλλοντος. Κυρία κυρία Ιώβα, ε, μέλος της ΣΥΤΡΕ. Κυρία Επίτροπε, ε, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, αγαπητή Σιλβή που έχουμε την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην προφορική σου δήλωση μίλησε για τι σημαντικότερε προκλήσει που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Η κοινή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική είναι κάτι που στόχο έχει την άρση των φραγμών της ενίας αγοράς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες να το συζητήσουμε και μεταξύ μας και γνωρίζω ότι είσαι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης της βιομηχανικής μας στρατηγικής. Συμφωνώ. Επίσης, θεωρώ ότι η προσέγγιση θα πρέπει να δράζεται στα ευρωπαϊκά συμφέροντα, θα πρέπει να είναι αμυγής ευρωπαϊκή και να μην ε, χωρίζει την Ευρώπη σε βορρά, νότο, ανατολή και δύση. Γνωρίζω από την εμπειρία σου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είσαι διαλλακτική, μπορείς να χτίσεις γέφυρες και να υλοποιήσεις συμβιβαστικέ λύσεις. Τι θα κάνεις στην επόμενη πενταετία στην βιομηχανική πολιτική, πώς θα βοηθήσεις τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από όποια χώρα και αν προέρχονται για να υποφεληθούν από την ενιαία αγορά και να είναι ανταγωνιστικές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Γκουλάρ, ευχαριστώ κύριε Διαβαλοβά, αγαπητή Μαρτίνα. Συνήθω μεταξύ μα μιλάμε Ιταλικά. Εν πάση περιπτώσει, θα αφήσουμε αυτό. Δυστυχώ δεν μιλάω τσεχικά. Ειλικρινά πιστεύω, έφυγε ο, ο άλλος συνάδελφος, όταν ε, λένε οι ευρωβουλευτέ ότι όλο γενικότητε μα λέτε, δεν λέτε τι θέλετε ακριβώ να κάνετε. Ναι, αλλά εγώ είμαι υπέρ τη συλλογική προσπάθεια, τη ομαδική προσπάθεια. Ε, και στο Κοινοβούλιο αυτό έκανα, όταν είχαμε ομάδα συγγητών ε, ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ίδιο θα κάνω. Θα λάβω υπόψη και τη γνώμη των συναδέλφων. Αν αρχίσουμε με πομπόδεις δηλώσεις και περνάμε σαν ηλίθιοι και δεν ευνοούμε το ομαδικό πνεύμα. Μιλήσατε για το χάσμα Ανατολής Δύσης. Είχα συνεργαστεί με τον Επίτροπο Πρόντι όταν ετοιμάζαμε τη διεύρυνση και ο κύριος Πρόντι ε, χαρακτήριζε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε την Επιτροπή της Διεύρυνσης και ήταν μια στιγμή πραγματικά πρωτοφανούς ευρωπαϊκής ε, αντάμωσης. Είχαμε την αίσθηση της ελευθερίας, της προόδου, είχαμε την Γερμανική Επανένωση που ήταν πραγματικά κάτι το καταπληκτικό που έγινε με ειρηνικό τρόπο. Ε, επίσης είχαμε και στην ε, Τσεχία ε, κορυφαίες προσωπικότητες όπως το Βάτσλα Χάβελ και τη Βελούδινη ε, Επανάσταση, την ανέμακτη μετάβαση. Και φυσικά ε, έχουμε μερικές φορές διαφωνίες, συζητούμε πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, τις δεξιότητες, αλλά θα πρέπει να περάσουμε αυτή τη σελίδα της αντιπαράθεσης. Και το είπα και προηγουμένως, αντιμετωπίζουμε ανταγωνισμό από τρίτες χώρες που έχει τεράστια μέσα, μεγάλη δύναμη, μερικές φορές δεν σέβεται τους κανόνες και δεν θα πρέπει να σκάβουμε το λάκκο μας ε, ενισχύοντας τον κατακαιρματισμό στη βιομηχανία, στον πολιτισμό, στο 5G, στην εσωτερική αγορά, σε όλους τους τομείς θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ε, ο κύριος Μπούζεκ φαντάζομαι ενδιαφέρεται για τη μετάβαση κάποιων ε, βιομηχανιών. Πιστεύω ότι θα ξαναβρούμε τις καλές συνήθειες της συνεργασίας μεταξύ μας. Κυρία Διαμπάλοβα, θέλετε να υποβάλλετε επερώτηση. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ευχαριστώ. Η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική σχετίζεται με την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, θα πρέπει όμως τα αποτελέσματα της έρευνας να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Μιλήσατε για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα ε, του Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης ε, και του οργανισμού GSA για τη διαχείρισή του που βρίσκεται στην Πράγα. Αυτό το πρόγραμμα, θα, αυτός ο οργανισμός θα μετατραπεί σε Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός. Και παρόλο που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα έχει ευρύτερο πεδίο αρμοδιοτήτων, ο προπολογισμό του είναι πενιχρός. Πώς θα καταφέρει ο οργανισμός να ανταπεξέλθει στην αποστολή του στη διαστημική πολιτική που είναι μία από τις ε, σημαντικές προκλήσεις του χαρτοφυλακίου σας. Η κυρία Γκουλάρ, ευχαριστώ που αναφερθήκατε στο διάστημα και στον οργανισμό που έχει έδρα την Πράγα, τον GSA. Είναι χαρακτηριστικό τομέα που δείχνει ότι αν κάνουμε καλέ επενδύσει και συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα, θα κρατήσουμε την τεχνολογική μα υπεροχή. Και το διάστημα έχει σημασία για τα μαζικά δεδομένα, για την πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα, το, το χρησιμοποιούμε καθημερινά στα smartphone μας. Βοηθάει τους γεωργούς να προβλέψουν καλύτερα ε, τον καιρό και να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό στις καλλιέργειές τους. Ο τομέας του διαστήματος είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, ο προϋπολογισμός του οργανισμού θα εξαρτηθεί από το ΠΔΠ, από το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελπίζω να είναι κατάλληλος για, για το έργο του. Ε, Έχουμε το θέμα της διακυβέρνησης του διαστήματος. Έχουμε επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος που βρίσκεται στο Παρίσι, που είναι διεθνής οργανισμός. Οπότε θα πρέπει όλους αυτούς τους φορείς διακυβέρνησης να τους ε, ε, κάνουμε να λειτουργήσουν καλά σε ένα περίπλοκο πλαίσιο. Οπότε θα φροντίσω όσο περνάει από το χέρι μου να έχει τα κατάλληλα μέσα και πόρους ε, ο οργανισμός αυτός. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ο ο κύριος Έλερ από την Επιτροπή Ήτρε και το ΕΛΚ. Κυρία Κουλάρ, τρεις ε, σημαντικές γενικές διευθύνσει ε, θα έχετε στα αρμοδιότητά σας, ε, την Connect, την Grow και τη Νέα για την Άμυνα. Αυτό ε, θα απαιτήσει ε, έναν θηλυκό Ηρακλή, είναι άνευ προηγουμένου. Ε, υπάρχουν τόσα θέματα, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, το Γαλιλαίο Κοπέρνικος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν πιστεύετε ότι οι κατηγορίες που πιθανότατα να αντιμετωπίσετε να είναι ασήκωτο βάρος για σας τελικά. Δεν νομίζετε ότι θα απαιτήσει το χρόνο σας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ασχοληθείτε με όλη αυτή την πολυπλοκότητα και οι ε, νομικές αυτές κατηγορίες που αντιμετωπίζετε και εύχομαι να μην είναι αλήθεια. Προσπαθώ να το πιστέψω κιόλα, αλλά δεν θεωρείτε ότι αυτός ο ακρογωνιός λήθος της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, απαιτεί όλη την προσοχή σας και τα θέματα αυτά δεν ε, τα έχουμε θίξει μόνο εμείς. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσετε σε όλα αυτά. Κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Πολλέ ερωτήσει τέθηκαν που πήγαιναν στην ίδια κατεύθυνση και έχετε κάθε δικαίωμα, διότι είστε εδώ για να διαπιστώσετε κατά πόσον ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σα μπορεί να αναλάβει την αποστολή που του ανατέθηκε ή τέλος πάντων θα ανατηθεί. Εγώ δεν θέλω να ισχυριστώ ότι είμαι superwoman. Σίγουρα πάντω ευκαιρίε όλοι αξίζουν. Αυτό το χαρτοφυλάκιο μου το ανέθεσε η κυρία Φοντερ Λάιεν και έχει κάποιε ελπίδε. Τώρα, συνολικά ε, είναι θέμα εξισορρόπηση των ε, αρμοδιοτήτων σε όλη την ε, Επιτροπή. Η κυρία Φεστάγκερ έχει την, ε, στον συντονισμό πολλών διαφορετικών τομέων, ο κύριο Ντομπρόφσκι το ίδιο. Ο καθένα στην Επιτροπή έχει πολλέ διαφορετικέ και ποικίλε αρμοδιότητε. Και εκτελεστική εκτελεστικοί αντιπρόεδροι μαζί με τον κύριο Τίμερμαν είναι ιδιαίτερα φορτωμένη με δουλειά. Εγώ δεν το μετανιώνω. Και όπω είπα και προηγουμένω, επειδή έχω βαθύ δεσμό Μάλλον, επειδή υπάρχει ε, σαφή διασύνδεση μεταξύ τη ψηφιοποίηση και τη ανάγκη μεταμόρφωση τη βιομηχανία μα, τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Βεβαίω θα στηριχθώ στι υπηρεσίε και του ε, συνεργάτε μου εδώ ε, και την λειτουργία ω κολεγίου των επιτρόπων. Όμω δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Έλερ. θέλουμε να είμαστε κινητήρια δύναμη. Θέλουμε να είμαστε αυτοί που θα φέρουν την πρωτοβουλία, τον ενθουσιασμό και την ορμή. Αλλά ο κ. Σπέν ήταν εδώ προηγουμένω, άλλοι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί μαζί μου. Ε, όταν κάναμε όλη τη μεταρρύθμιση με τον κύριο Μπάλ, α πούμε, ναι, τη μεταρρύθμιση των χρηματοοικονομικών. Πολύ βαρύ, πολύ δύσκολο, ε, μέσω χρηματοοικονομική κρίση. Επί χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα. Και με την ε, light touch κάτι κάναμε. Εδώ λοιπόν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω περισσότερε ε, ικανότητε από του άλλου άλλου. 24 ώρο ζω και εγώ τη μέρα. Προσπαθώ να το αξιοποιήσω το καλύτερα δίνει, αλλά όπω ε, έχει πει μια μεγάλη κυρία τη Γερμανία, κύριε Έλλερ, διασάφεντα. Θα τα καταφέρουμε. Η επερώτησή σα. Όχι, ευχαριστώ, δεν έχω. So, uh, thank you very much, uh, colleagues, for your questions. Ε, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα θα έχει πάλι η κυρία Γκουλάρ, αν το επιθυμεί, ένα πεντάλεπτο για τα καταληκτικά της σχόλια. Παρακαλώ, κυρία Γκουλάρ. Κύριε Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ και αγαπητό κοινό, αν έχει ακόμη το κοινό την υπομονή και μας παρακολουθεί ακόμη. Θα ήθελα μετά τη σημερινή συζήτηση να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, οι δημόσιες αυτές ακροάσεις είναι ε, μια άσκηση δημοκρατίας, νομίζω. Δεν υπάρχει στα πολιτικά μας συστήματα κάτι αντίστοιχο πριν την ανάληψη ε, ενός αξιώματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα το δημοκρατικό και η συζήτηση έμεινε σε ευγενικά επίπεδα παρά τη διαφορά απόψεων και την αντιπαράθεση που υπάρχει μερικές φορές και έδειξε η συζήτηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εργάζεται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζω ότι ε, θα αξιολογήσετε ένα άνθρωπο με την πορεία του, με τα λάθη του. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που με κάνουν υπαρήφανη, αλλά που ίσως για το οποία έχω μετανιώσει. Επίσης, ε, ελπίζω να διαβεβαιωθήκατε για την ακαιρεότητά μου, ε, γιατί είμαστε όντως θεματοφύλακες της σωστής χρήσης των ε, κονδυλίων των φορολογουμένων, εννοείται. Και έχετε δίκιο που απαιτείται αυτόν τον έλεγχο. Σας έδωσα κάποιες εγγυήσεις ε, και δικαστικές και πρακτικές και κυρίως σας επισήμενα το τεκμήριο της αθωότητας που κατοχυρώνεται σε πολλούς χάρτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι είναι από τις αξίες που μας ενώνουν. Και αν αποφασίσετε τελικά να μου δώσετε την έγκρισή σας, θα προσπαθήσω να υπηρετώ την ευρωπαϊκή ιδέα, όπως έχω κάνει τα τελευταία 30 χρόνια, σε διαφορετικούς φορείς, με διαφορετικό κόσμο, αλλά με ένα και μόνο στόχο, την εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Και ξέρετε, πριν την ανάληψη των καθηκόντων, οι επίτροποι πηγαίνουν στο δικαστήριο και δίνουν όρκο. Ε, δίνουν υπόσχεση ε, πίστης, ανεξαρτησίας, αμεροληψίας. Και αν μου δώσετε την ευκαιρία να το κάνω, ε, σας διαβεβαιώ ότι θα σας υπόσχομαι να τηρήσω όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία. Και τέλος, ήθελα να σας πω ότι οι ερωτήσεις που θέσατε και που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ε, με οδηγούν στη σκέψη ότι η αποστολή της Επιτροπής θα είναι πολύ δύσκολη και απαιτητική. Όπως είπε ο κύριος Μπομπάρ, έχουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στον άνθρακα, στην κατανάλωση, σε ένα συγκεκριμένο είδος διαβίωσης, μετακίνησης, παραγωγής και όλα αυτά αμφισβητούνται από τις κλιματικές αλλαγές και από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Επίσης, είμαστε, και ας μην το ξεχνάμε, οι προνομιούχοι του πλανήτη για δεκαετίες και για αιώνες είχαμε την υπεροχή και την κυριαρχία και την ασκούσαμε μέρημνα. Η κατάσταση όμως έχει αλλάξει και γεωπολιτικά και δημογραφικά και όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο πια ζωής μας. Επίσης, αν με, με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, θα διευκολύνω τη ρηξικέλευθη μεταμόρφωση που μας περιμένει και θα την προσεγγίσω με ταπεινοφροσύνη και με τριοφροσύνη. Γενικώ, ε, εσείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είστε κινητήρια δύναμη της ολοκλήρωσης, γιατί η κυβερνήση είναι πολύ πιο κοντά σε τοπικά κριτήρια και είναι πιο διστακτική ε, απέναντι σε μια συνολική θεώρηση. Οπότε, σε έναν ε, επικίνδυνο κόσμο που αφισβητούνται η, πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, ε, η, συμφωνία για το κλίμα, σε έναν κόσμο που είναι λιγότερο συνεργατικός και που ίσως ε, φαίνεται πιο επικίνδυνος από ό,τι σκεφτόμαστε στο παρελθόν, σε έναν κόσμο που ο πολιτισμός δεν έχει την θέση που το αξίζει, δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις, θα πρέπει να ανασκουμποθούμε και να περάσουμε στο έργο. Ω Ευρωβουλευτής προσπάθησα να, περάσω, να ξεπεράσω τα σύνορα, τα κομματικά, τα εθνικά, τα πνευματικά μεταξύ Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότου, όλα όσα μα επιβάρυναν τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσω σε αυτή την προσπάθεια να ξεπερνάω τα σύνορα. Και επίση, ε, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να βρουν γέφυρες μεταξύ τους. Δεν είναι άνθρωποι που θέλουν την αντιπαράθεση. Η Ευρώπη είναι διάλογος και συμβιβασμός και είναι ικανότητα να πει κανείς δεν θα κερδίσω 100% θα κάνω κάποιε υποχωρήσεις αλλά το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο σε συνεργασία παρά ο καθένας μόνος του. Ο Ζαμονέ είπε ε, εμείς ενώνουμε τους ανθρώπους, δεν συνασπίζουμε τα κράτη. Αυτό ήθελε να κάνει η Ursula von der Leyen, να ενώσει τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Μαζί με τους άλλους ε, επιτρόπους αυτό θα κάνω, αν ε, με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ. Uh, Λίγα λόγια τώρα από την κυρία Τεσούτερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οριστήσα Επίτροπο για τις απαντήσεις της και που συμμετείχε στη συζήτηση αυτή με τις δύο επιτροπές μας. Ε, το χαρτοφυλάκιο σας περιέχει πολλά θέματα, γι' αυτό ε, χρειάστηκε να οργανώσουμε την ε, συνεδρίαση αυτή με αρκετές επιτροπές και θα ήθελα να πω ότι χάρη στην εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές ε, ήταν ε, πολύ καλή ε, διοργάνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συμπρόεδρό μου, την κυρία Βαλεάν, καθώς και τους πρόεδρους των επιτροπών Καλτ και Γιούρι που συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Και θα κλείσω δίνοντας το λόγο πάλι στην κυρία Βαλεάν και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην ε, διοργάνωση αυτή. Ε, τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Ε, θα έχουμε μία συνάντηση των συντονιστών των δύο επιτροπών, Ήτρε και Ίμκο, για να αξιολογήσουμε τις απαντήσεις της οριστής σας επιτρόπου. Θα εξετάσουμε τις, τα γενικά προσόντα και την ε, ανεξαρτησία και την ε, καταλληλότητα για